Καλησπέρα αγαπητοί συνάδελφοι. Ας αρχίσουμε τη συνεδρίαση της Επιτροπής μας. Πρώτα απ' όλα, η μερίσια διάταξη. Υπάρχουν σχόλια. Παρακαλώ. Με η κυρία Μπιόρκ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Από την ομάδα μας στείλαμε ένα mail από την GUE-NGL να αναβληθεί η σημερινή ψηφοφορία για την ερώτηση και το σχέδιο ψηφίσματος όσον αφορά τον ρόλο των γυναικών. Υπάρχουν πάρα πολλές ανησυχίες από την πλευρά μας και θα σας πω γιατί. Έχουμε συναντηθεί με την κοινωνία των πολιτών και μας έχουν εκφράσει την ανησυχία τους και διάφορες ομάδες μάλιστα τις οποίες κανονικά εξυπηρετεί αυτό το κείμενο δεν τους ικανοποιεί αυτό το κείμενο. Εκφράζουν ανησυχίες. Ε, αυτό πρέπει να μας τυπεί στο καμπανάκι του κινδύνου. Οι ομάδες κατά του ρατσισμού, οι ομάδες υπέρ των δικαιωμάτων της γυναίκας λένε ότι στιγματίζονται συγκεκριμένες ε, ομάδες, όπως οι γυναίκες μετανάστριες, και είναι ε, σαφές από τη δουλειά που έχω κάνει εγώ με τους συναδέρφους από άλλες πολιτικές ομάδες και για άλλες μορφές ε, ακραίων τάσεων άκρας δεξιάς ή οτιδήποτε. Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί δεν θέλει να μιλήσει για αυτά ο συγητή, Εγώ το νιώθω στο πετσί μου ότι πρόκειται για απειλή. Εγώ δεν νομίζω ότι είμαστε αξιόπιστοι εάν ε, ετοιμάσουμε ένα κείμενο που δεν λαμβάνει υπόψη του αυτές τις ακροδεξιές τάσεις. Είναι θέμα λοιπόν υπευθυνότητα, είναι θέμα κοινοτήτων και εγώ πιστεύω ότι αυτό το κείμενο μπορεί να βελτιωθεί, να είναι ικανοποιητικό και εξυπηρετικό και για την κοινωνία των πολιτών και για μας τους ευρωβουλευτές, αλλά να μην πιέσουμε τα πράγματα να περάσει σήμερα έτσι. 2 Απριλίου, αν το εγκρίνουμε, που αυτό επιλέγουμε εμείς, μια χαρά θα είναι. Αυτό προτείνω λοιπόν στην Επιτροπή μας να αναβληθεί η ψηφοφορία και να γίνει στις 2 Απριλίου. Ευχαριστούμε κύριε Βιώνο. Κύριε Σουρτασούν. Εγώ θέλω να στηρίξω το αίτημα της ΓΚΟΕ NGL. Και εγώ βλέπω ότι δεν φαίνεται να είμαστε έτοιμοι για να ψηφίσουμε αυτή την έκθεση. Και θα κάνει κακό στην εικόνα της Επιτροπής μας τώρα που βρισκόμαστε στο τέλος της θητείας αν εγκρίνουμε αυτή την έκθεση έχοντας προηγουμένως λάβει πολύ συγκεκριμένες ανησυχίες που έχουν εκφράσει οι διάφορες μη κυβερνητικέ οργανώσεις όπως το δίκτυο κατά του ρατσισμού συμφωνούμε ότι το ψήφισμα αυτό θα ψηφιστεί μόνο στην Επιτροπή μας, έτσι, όχι στην Ολομέλεια, οπότε έχουμε χρόνο. Γι' αυτό ζητούμε και εμείς να καθίσουμε πάλι να διαπραγματευτούμε, ώστε να καθησυχαστούν οι διάφορες ανησυχίες. Δώστε μας λίγο περισσότερο χρόνο πριν φτάσουμε στην ψηφοφορία. Ευχαριστούμε κύριε Ρουτασούν. Χτες ενημερώθηκα από τους συντονιστές ε, της ομάδας Γκουε και των Πρασίνων ότι θέλουν να αναβληθεί η ψηφοφορία της προφορικής ερώτησης και του ψηφίσματος για το ρόλο των γυναικών στην ε, πρόληψη της ε, ριζοσπαστικοποίησης. Βασιζόμαστε στο άρθρο 109 του κανονισμού. Η πρόταση για αναβολή θα ψηφιστεί στην αρχή των ψηφοφοριών που έχουμε σήμερα. Στις 5 δηλαδή θα ψηφίσουμε για αυτό το αίτημά σας. Παρακαλώ εσείς. Ευχαριστώ. Είμαι σκιώδης από τους σοσιαλιστές και στηρίζω και εγώ αυτό το αίτημα. Ε, πιστεύω και εγώ ότι έχει βάσει αυτό που λένε η ριζοσπαστικοποίηση. Ε, συχνά είναι ε, θέμα ε, παρεξηγήσεων. Είναι κάτι που με απασχολούν πάρα πολύ. Βλέπετε είμαι και εγώ από μια περιοχή με πολλές και διαφορετικές προελεύσεις του κόσμου, με πολλούς μουσουλμάνους και βλέπω ότι οι γυναίκες, τα παιδιά πολύ συχνά είναι θύματα της Ισλαμοφοβίας και κάτι το οποίο μάλιστα επεκτείνεται σε ολόκληρη την Ευρώπη. Οπότε, ναι, θέλω να υπάρχει αυτή η έκθεση, αλλά να είναι ισορροπημένη. Και εγώ έχω ανησυχίε για το κείμενο όσο έχει τώρα. Έχουμε συνεργαστεί συχνά μαζί. Πιστεύω και εγώ ότι οι γυναίκες έχουν ρόλο να παίξουν, αλλά δεν βοηθάει να στιγματίζουμε τη μία ή την άλλη ομάδα ανθρώπων. Ευχαριστώ. Παρακαλώ εσείς. Εγώ είμαι κατά τη αναβολή τη ψηφοφορία. Εγώ καταλαβαίνω ότι όταν αρχίσουμε τι ψηφοφορίε, τότε θα ψηφίσουμε και θα αποφασίσουμε τι θα κάνουμε. Αλλά σα λέω ότι εγώ πιστεύω ότι έχει ολοκληρωθεί η συζήτηση. Σίγουρα υπάρχουν κάποιες απόψεις διαφορετικές. Υπάρχει κόσμος που δεν συμφωνεί και δεν θα συμφωνήσει. Η συζήτηση αυτή για μένα έχει ολοκληρωθεί. Ας ψηφίσουμε και να κλείσει ο φάκελος. Αυτή είναι η δικιά μου γνώμη. σε ευχαριστούμε. Άλλα σχόλια. Όχι, ωραία. Θα ψηφίσουμε λοιπόν στις 5 σήμερα το απόγευμα. Δεν υπάρχουν άλλα σχόλια. Εντάξει. Οπότε έγκρινεται η μερίσια διάταξη. Δεύτερο σημείο στην ημερήσια διάταξη. Έγκριση των πρακτικών τη 8η Νοεμβρίου και τη 21η Νοεμβρίου επίση. Αν δεν υπάρχουν σχόλια για τα πρακτικά, θεωρούνται εγκεκριμένα. Ανακοινώσει τη Προέδρου. 3.1. Στη συνάντηση της 23 η Ιανουαρίου, οι συντονιστέ αποφάσισαν να ακυρώσουν την αποστολή στη Γερμανία που είχε σχεδιαστεί για τα τέλη αυτού του μήνα αρχικά. Με γραπτή διαδικασία, ε, στις 21 Φεβρουαρίου, αποφάσισαν οι συντονιστέ να εγκρίνουν πρωτοβουλίε των ε, σύν εισηγητών όσον αφορά την πρόσβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην σύμβαση της Κωνσταντινούπολης. Πρόκειται για την κυρία Κοράτσα Μπίλτ και την κυρία Ρεβό Νταλόν Μπονφουά και ζητούν την γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για την επιλογή της κατάλληλης νομικής βάσης για την απόφαση και για την υπογραφή των συμπερασμάτων και μιλάει για δύο διαφορετικές υπογραφές και για την λογοδοσία της πρακτικής μια κοινή συμφωνίας από το Συμβούλιο στις αποφάσεις του και για την εφαρμογή της αρχής της ειλικρινούς συνεργασίας υπό το φως του εκπεφρασμένου στόχου στην Ευρωπαϊκή Ένωση να ολοκληρώσει και να συνυπογράψει τη σύμβαση. Για τον ίδιο φάκελο αποφάσισαν οι συντονιστέ να στείλουν επιστολή στην Ρουμανική Προεδρία σχετικά με την ε, απόφαση των συμπερασμάτων για την ε, προσχώρηση στο Συμβούλιο. Θέλω επίσης να καλωσορίσω εδώ διάφορες ομάδες επισκεπτών που θα βρίσκονται εδώ στη συνεδρίασή μα. Η κυρία Ζωάννα πρώτα απ' όλα έχει επισκέπτες από την Οργάνωση Γυναικών ε, του Σοσιαλιστικού και Δημοκρατικού Κόμματος της Ρουμανίας. Η κυρία Βόζεμπερκ κάλεσε μια ομάδα φοιτητών αγγλικής φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Και η κυρία Πετήρ θα έχει προσκεκλημένους από την Κροατία. Πρόκειται για την Ένωση Πιο Υποχρηματικές ε, Γυναίκες της Κροατίας. Και δημοσιογράφοι επίσης όταν θα ψηφίσουμε ε, την γνωμοδότηση για τη CIP. Οι δημοσιογράφοι θα μαγνητοσκοπήσουν κομμάτια της ε, συνεδρίασης. Συνεχίζουμε, σημείο 4. Η ισότητα μεταξύ των δύο φίλων στη Γεωργία. Έχουμε ανταλλαγή απόψεων. Η ε, κυρία Ματσοκοσφίλη είναι η συγγήτριά μας εδώ, η ομιλήτριά μας. Θα μας μιλήσει για ανταλλαγή. Θα έχουμε συζήτηση μεταξύ μας και έτσι θα ενημερωθούμε για το τι δουλειά έχει γίνει τα τελευταία χρόνια και θα συζητήσουμε παρετέρω δράσεις και προκλήσεις. Θα σας δώσω το λόγο στην κυρία Μαρτσεσβίλη που είναι η πρόεδρος του Κοινοβουλίου της Γεωργίας. Παρακαλώ έχετε το λόγο.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 Ευχαριστώ πολύ. Κυρίε και κύριοι, αγαπητοί προσκεκλημένοι, ευχαριστώ πολύ για αυτή τη δυνατότητα να σας απευθύνω το λόγο και να σας παρουσιάσω τις εξελίξεις για την ισότητα του φίλου στην Γεωργία. Πριν περάσω στην ουσία της συζήτησης, θέλω να σας πω γιατί θελήσαμε τόσο πολύ να διοργανωθεί αυτή η ακρόαση και το Κοινοβούλιο να ακούσει τι πρόοδο έχει επιτελεστεί στην Γεωργία. Έχουμε κάνει μεγάλη πρόοδο. Έχουμε πετύχει σημαντικά αποτελέσματα με σημαντικές προκλήσεις και μέχρι τώρα είχαμε σοβαρή στήριξη από το Κοινοβούλιο, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και χωρί όλη αυτή τη στήριξη νομίζω ότι η χώρα μου δεν ε, θα μπορούσε να ξεπεράσει τι δυσκολίε που ξεπέρασε. Ήθελα λοιπόν να σα ευχαριστήσω για την ευκαιρία και να χρησιμοποιήσω τον χρόνο που μου δίνετε για να σα πω τι καταφέρατε να πετύχουμε εμεί ή τι εμεί πετύχαμε χάρη στη δική σα παρέμβαση για την ε, μάχη υπέρ τη ισότητα των φύλων στην Γεωργία και για τα αποτελέσματα που εντό μικρού χρονικού διαστήματος ε, καταφέραμε να πετύχουμε με πολύ πάθος, ζήλο και ενθουσιασμό. Σας ευχαριστούμε λοιπόν πολύ. Ευχαριστούμε πολύ για τη βοήθεια της Ευρώπης λοιπόν και του Ευρωκοινοβουλίου. Με το Ευρωκοινοβούλιο Βλέπω ότι κάποιοι βρίσκονται εδώ, οι Κλέρ βρίσκεται εδώ. Ε, με κάποιους από τους βουλευτές, το κοινοβούλιο έχει πολύ στενή, ε, εμείς έχουμε πολύ στενή συνεργασία. Ε, πολύ καλή επικοινωνία που είναι κέρια σημασία. Η σχέση μας είναι πολύτιμη και ελπίζουμε να συνεχιστεί. Όσο για τις βασικές πτυχές της ισότητας του φίλου στην Γεωργία, να αναφερθώ στους βασικότερους τομείς. Θα προσπαθήσω να μην μπω στις ε, λεπτομέρειες για να εξοικονομήσουμε χρόνο και να έχουμε περισσότερο χρόνο για το Q&A, τις ερωταπαντήσεις, αλλά οι σημαντικότερες πτυχές. Θα σχολιάσω πέντε βασικές κατευθύνσεις. Πρώτα απ' όλα η βία λόγω του φύλου, δεύτερον η διακριτική μεταχείριση κατά των γυναικών, τρίτον η συμμετοχή των γυναικών στα πολιτικά πράγματα, θα σας πω που έχουμε φτάσει και ποια πρόοδος έχει επιτελεστεί. Μετά η οικονομική ε, χειραφέτηση των γυναικών, σημαντικό μέρος της δουλειάς μας και τελευταίο και όχι, σημαντικό, και όχι λιγότερο σημαντικό, η ενίσχυση των θεσμών που δημιουργούνται ή έχουν δημιουργηθεί. Και εκεί θέλουμε να υπάρχει η ισότητα των φύλων που να εκφράζεται στη λειτουργία τους. Αυτές είναι οι πέντε βασικές κατευθύνσεις που θα ακολουθήσω στην ομιλία μου. Όπως υπόθηκε στην αρχή, θα σας παρουσιάσω το Κοινοβούλιο της Γεωργίας. Είμαι βουλευτής, είμαι πρόεδρος της Επιτροπής για την Ισότητα των Φίλων στο Γεωργιανό Κοινοβούλιο και βεβαίως εκεί συμμετέχουν διαφορετικές πολιτικές ομάδες, όπως φανταστήκατε οι πολιτικές ομάδες που βρίσκονται στο κοινοβούλιο μας, όλες εκπροσωπούνται και στο δικό μας Συμβούλιο Επιτροπή για την Ισότητα των φίλων. δουλειά είναι να συντονίζουμε τις προσπάθειες και να προωθούμε την ατζέντα για την ισότητα των φύλων στην Εθνική Βουλή. Η δουλειά μας έχει εγκομιαστεί ε, επανειλημμένως τα τελευταία δύο χρόνια. Και νομίζω ότι είναι μια καλή ευκαιρία, μια ακόμα καλή ευκαιρία, για να σας πούμε τι κάνουμε και ποιες είναι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε. Καταρχάς, η έμφυλη βία, όπως ονομάζεται, η βία βάση του φύλου. Μια, ε, ένα πρόβλημα που έχει αντιμετωπίσει πολλά χρόνια η χώρα μας την έχει ταλανίσει. Όπως φαντάζεστε, επί πολύ καιρό υπήρχε πρόβλημα με την βία λόγω του φίλου. Το βασικό πρόβλημα ήταν η ευαισθητοποίηση και η νοοτροπία που επικρατούσε στην κοινωνία γενικότερα. Θεωρούσαν ότι η ενδοοικογενειακή βία και η βία στα πλαίσια της οικογένειας ήταν θέμα ιδιωτικό. Έπρεπε να μείνει κρυφό. Τα ενίκομοι ενδύμου αυτό αντικατοπτρίζεται και στην ε, δουλειά των θεσμικών φορέων. Όταν τα θύματα λόγω χάρη τηλεφωνούσαν στην αστυνομία, η αστυνομία ε, δεν έμπαινε και κατευθείαν ε, στο προσκήνιο για να προστατεύσει το θύμα. Πριν από δύο χρόνια όμως κυρώσαμε την σύμβαση της Κωνσταντινούπολης. Ένα σημαντικό έγγραφο και με την κύρωσή της εγκρίναμε και τροποποιήσαμε τουλάχιστον ε, καμιά εικοσαριά νόμους σχέση με το θέμα αυτό. Με αυστηρότερους λοιπόν κανόνες στην νομοθεσία μας πλέον για την προστασία των θυμάτων και κατά των ε, δραστών. Πριν εγκρίνουμε την σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, είχαμε κάποια νομοσχέδια και νόμους που εγκρίθηκαν, αλλά το βασικό ε, εργαλείο που έλειπε ήταν αυτό τη υλοποίηση τη εφαρμογή. Αυτό που διασφάλιζε ότι όλοι οι κανόνε που έχουμε, όλοι οι κανονισμοί κατά τη ενδοοικογενειακή, τη έφυλη βία, ότι αυτά θα εφαρμόζονται. Σε συνδυασμό με την κύρωση τη Σύμβαση τη Κωνσταντινούπολη, λοιπόν, και τι ε, τροπολογίε τη, κάτι που κάναμε και που έχει αποδώσει είναι ότι δημιουργήσαμε υπηρεσία ειδική για τα ανθρώπινα δικαιώματα εντός του Υπουργείου Εξωτερικών ένα πολύ καλό εργαλείο που εργάζονται κάτι υπέροχες γυναίκες και ασχολούνται με την παρακολούθηση της ε, διαδικασίας, ε, όποια έκθεση ή αναφορά ή καταγγελία ή μήνυση φτάνει στα χέρια του Υπουργείου Εσωτερικών, όχι Εξωτερικών για καταγγελία ενδοκογενειακής ή εμφύλης βίας ε, κοιτάζουν ότι είναι ποιότητας και περιεχομένου και ότι υπάρχει απαραίτητη εξακολούθηση και συνέχιση έρευνα στην κάθε υπόθεση. Έχουμε θαυμάσει αποτελέσματα. Για να σας δώσω στοιχεία, το 2014 αριθμό αριθμός διώξεων κατά των δραστών έμφυλης βίας, ο συνολικός αριθμός ήταν 550 υποθέσεις. Πέρσι ο αριθμός πήγε τις 3.050. Εξαπλασιασμός ε, πέρσι σε σχέση με το 2014. Η αριθμητική αυτή αύξηση σημαίνει ότι αυξήθηκε βέβαια και το ποσοστό εγκληματικής ε, δράσεις. Αλλά δεν ήταν ότι διαπράχθηκαν περισσότερα εγκλήματα. Αποκαλύφθηκαν περισσότερα, καταγγέλθηκαν περισσότερα. Κατά των ανδρών, εντός της οικογένειας, εκτός οικογένειας. Ε, αυτά που δεν καταγράφονταν πουθενά και ε, παρέμεναν σε πλήρη ατιμορρησία. Με τους νέους αυτούς κανόνες, με τους νέους νόμους και μηχανισμούς που εφαρμόσαμε, είχαμε δραματική αλλαγή. Επιπλέον, κάτι άλλο που άλλαξε Άρδιν είναι ότι το κράτος άρχισε να χρησιμοποιεί σοβαρότατα ασφαλιστικά μέτρα κατά των δραστών. Τα μη ασφαλιστικά μέτρα που χρησιμοποιούνταν προηγουμένως στις περισσότερες υποθέσεις Ακόμη και αν το θύμα τηλεφωνούσε στην αστυνομία, ε, δεν έδιναν τίποτα ως αποτέλεσμα. Ο δράστη ξέφευγε με καμιά ε, σύντομη εκδίκαση τη υπόθεσή του στο δικαστήριο χωρίς ποινική διάσταση. Τώρα όμως χρησιμοποιούμε πραγματικά ασφαλιστικά μέτρα με ποινικέ κατηγορίες κατά των δραστών. Επιπλέον ξεκινήσαμε να χρησιμοποιούμε τα προγράμματα διαχείρισης κινδύνου. Τι θα πει αυτό όπως και σε άλλες χώρες έχουμε τις περιπτώσεις γυναικοκτονιών, δολοφονίας γυναικών. Είναι περιπτώσεις έμφυλης βίας όπου φτάνουν σε ακραίο αποτέλεσμα, δηλαδή το φόνο της γυναίκας. Έχουμε πολλές τέτοιες περιπτώσεις γυναικοκτονίας. Ε, ε, εισαγάγαμε λοιπόν ένα σύστημα που ε, επιτρέπει να παρακολουθούμε τους δράστες, τους αυτούργους, πριν καταλήξουν στο δυστυχές αυτό αποτέλεσμα. Έτσι έχουμε περιορίσει τον κίνδυνο στο δυνατόν περισσότερο. Αυτό έχει εφαρμοστεί και έχει επιτρέψει να μειωθεί ο ρυθμός δολοφονίας γυναικών στη Γεωργία. Θα περάσω στη διακριτική μεταχείριση και τη σεξουαλική παρενόχληση, που είναι και το ζουμί της παρουσίασής μου. Η σεξουαλική παρενόχληση δεν ε, ρυθμίζεται νομοθετικό στη Γεωργία καθόλου. Αυτό στη δική μας την νομοθεσία δεν αντικατοπτριζόταν επαρκώς. Δεν υπήρχε καν ορισμός. Ήταν περισσότερο μέρος Μια σύσταση δικαστηρίου που την είχε ενισχύσει και, το, και η υπηρεσία του ανθρώπινου διαμεσολαβητή ήταν γενικώ διακριτική μεταχείριση. Αλλά η σεξουαλική παρενόχληση δεν ήταν αντικείμενο συγκεκριμένου ορισμού στην νομοθεσία μα. Όμω, με τη δουλειά του Συμβούλου για την Ισότητα των Φίλων στη Βουλή μα, και γενικότερα όμω έκανε το Κοινοβουλίο μα, εισαγάγαμε ένα πολύ σημαντικό νόμο που θα εγκριθεί στη Βουλή της χώρας και δίνει ένα λεπτομερέστατο διεξοδικό ορισμό για την σεξουαλική παρενόχληση. Ε, και προβλέπει μάλιστα και συγκεκριμένα εργαλεία και μηχανισμό για να προστατευτούν οι γυναίκε θύματα σεξουαλική παρενόχληση. Και πώ πρέπει να αντιδράσουμε σε περίπτωση που κάτι τέτοιο συμβεί. Αυτά έχουν καταρτιστεί σε πολύ καλή συνεργασία με εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών, τις οργανώσεις τους. Τους ευχαριστώ πολύ γιατί ήταν πολύ δραστήριοι, πολύ ενεργοί. Μας ε, διευκόλυναν στο Βουλή της χώρας για να εκπονήσουμε ε, το σωστό νομοσχέδιο. Πολύ σύντομα λοιπόν η Γεωργία θα έχει αυτό το ενισχυμένο πλαίσιο. Ένα βελτιωμένο νόμο κατά της διακριτική μεταχείρισης, για την καταπολέμηση κάθε μορφής αυτής και νέους κανόνες για την καταπολέμηση της σεξουαλικής παρενόχλησης. Θα είναι ένα μεγάλο βήμα πρόοδο αυτό, διότι επί χρόνια οι οργανώσεις γυναικείων δικαιωμάτων πίεζαν επιτέλους αυτό να περάσει. Το επόμενο θέμα της παρουσιασή μου είναι η συμμετοχή των γυναικών στα πολιτικά πράγματα. Εδώ απομένει ακόμα πολλή δουλειά. Υπάρχει τεράστιο περιθώριο βελτίωσης. Φέτο, η Γεωργία γιορτάζει 100 χρόνια ε, δημοκρατικού ε, πολιτεύματος. Βέβαια διέρχεσε πολύ λίγο λόγω της σοβιετικής κατοχής τότε, όμως πριν από 100 χρόνια η Γεωργία όχι μόνο δικαιώματα για τι γυναίκε που έβλεπε, αλλά είχε και γυναίκες βουλευτίνες οι οποίες ήταν ε, πολύ δραστηριές και έκαναν τεράστια δουλειά. Τότε λοιπόν η Γεωργία ήταν ήδη πολύ ευρωπαϊκή χώρα, στραμμένη προς την ευρωπαϊκή κουλτούρα. Όμως με τη ρωσική κατοχή έχασε πολλά. Και αφού ανακτήσαμε την ανεξαρτησία μας, ξεκινήσαμε από πάρα πάρα πολύ χαμηλό επίπεδο και ποσοστό παρουσίας των γυναικών στην πολιτική, και στι θέσει λήψη αποφάσεων. Εννέα μόνο γυναίκες στη Βουλή μας στην αρχή. Και δεν αυξήθηκε για πολύ αυτό ο αριθμό μέχρι σήμερα. Τώρα το ποσοστό γυναικών στη Βουλή είναι 15%. Απέχει πόρο από το να θεωρηθεί οκ ή τέλο πάντων αρκετό. Αλλά είναι και ένα πράγμα για το οποίο καμαρώνουμε. Η Γεωργία είναι η πρώτη χώρα στην όλη γεωγραφική περιοχή που προσφάτω τις περσινές εκλογές εξέλεξε την πρώτη γυναίκα πρόεδρο. Και αυτό είναι πολύ, δεν είναι ευκαταφρόνητο, όχι μόνο για τη δική μα τη χώρα, αλλά και για τις γειτονικέ. Καμία χώρα ε, στην περιοχή ε, της Κασπίας και του Καυκάσου δεν είχε γυναίκα πρόεδρο. Πέραν τι εκλογικέ διαδικασίε που χρειάστηκε να περάσει, όπω όλε οι γυναίκε, κατάφερε και να κερδίσει η γυναίκα αυτή. Ε, είναι μια γυναίκα που μπορεί να βοηθήσει στην αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στα πολιτικά πράγματα και στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σε κρίσιμες θέσεις και πόστα. Έχουμε πάνω από 25% γυναίκες ε, στην κυβέρνηση πλέον και Όπω σα είπα, 15% εκπροσώπηση γυναικών στη Βουλή εν γέννη. Όμω, αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι ότι όλε οι γυναίκε που είναι στη Βουλή έχουν πολύ σοβαρά χαρτοφυλάκια, βρίσκονται σε πόστα σημαντικά για την λήψη αποφάσεων. Έχουμε δύο αντιπροέδρου στη Βουλή, γυναίκε, τέσσερι προέδρου σημαντικότατων επιτροπών στη Βουλή, οκτώ αντιπροεδρου των επιτροπών, δύο επικεφαλεί πολιτικών ομάδων. Άρα είναι μικρό αριθμό των γυναικών, αλλά όλε είναι σε θέσει κλειδιά. Ε, κάνουν πολύ σοβαρή δουλειά στη Βουλή μα και αυτό είναι ένα θετικό στοιχείο και αποδεικνύει ότι χρειάζονται και άλλε. Θέλουμε περισσότερε από ό,τι έχουμε τώρα. Στο Συμβούλιο για την Ισότητα των Φίλων, στην Βουλή θέλουμε να υπάρξουν υποχρεωτικέ ποσοστώσει ε, για τη συμμετοχή των γυναικών. Είναι λίγο αμφιλεγόμενο θέμα αυτό και λίγο αντιφατικό ως εργαλείο, αλλά είναι αποτελεσματικό κιόλα για να υπερπηδήσουμε αυτό το πρόβλημα. Τη συμμετοχή των γυναικών στα πολιτικά πράγματα και σε σύντομο χρονικό διάστημα, μάλιστα. Επιτρέπει την αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στα πολιτικά πράγματα. Επίσης και ο εκλογικό μας νόμος, το σύστημα ε, περιμένουμε να αλλάξει για να επιτρέψει την συμμετοχή των γυναικών και στις εκλογές. Οι υποχρεωτικές ποσοστώσεις ψηφίστηκαν πέρσι στη Βουλή μας, αλλά δεν πέρασαν. Για εννέα μόνο ψήφους διαφορά. Πολύ κοντά ήταν ε, για να περάσουν. Έχουμε όμως 80% άνδρες που δεν είναι καθόλου, καθόλου διατεθειμένοι να εγκαταλείψουν το πόστο τους για να μπουν οι γυναίκες στην πολιτική. Δεν απλό λοιπόν να τους εκτοπίσουμε ή τέλος πάντων να τους πείσουμε. Έτσι δεν πέρασε ο νόμος, αλλά δεν το βάνουμε κάτω. Δεν παραδεινόμαστε, θα ξαναπιέσουμε να περάσει το νομοσχέδιο θα το ξαναυποβάλουμε και θα προσπαθήσουμε να συγκεντρώσουμε στήριξη για την πρωτοβουλία μας. Αυτή τη φορά μπορεί και να περάσει το νομοσχέδιο. Είναι σημαντικότατη πτυχή της δουλειάς μας. Το επόμενο θέμα που θέλω να αναπτύξω είναι η οικονομική χειραφέτηση των γυναικών. Και πάλι πρόκειται για έναν τομέα όπου χρειάζεται να γίνει πολλή δουλειά. Δυστυχώ έχουμε τεράστιο μισθολογικό χάσμα. Οι άντρε και οι γυναίκε λαμβάνουν διαφορετικού μισθού για την ίδια δουλειά. Το Συμβούλιο Ισότητας των Φίλων στο Κοινοβουλίο έχει δώσει προτεραιότητα στη χειραφέτηση των γυναικών, τουλάχιστον για τη φετινή χρονιά. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να διευκολύνουμε τη δημιουργία εργαλείων και μηχανισμών ώστε να χειραφετηθούν κι άλλο οικονομικώς οι γυναίκες. Ε, ανανεώνουμε και αναθεωρούμε τον κώδικα τον εργασιακό μας για να μπορούν οι γυναίκες να απασχολούνται, να είναι εργοδότριες και να έχουν την οικονομική τους αντεξαρτησία ευκολότερα. Θα ε, προσαρμόσουμε και τα προγράμματα κρατικής βοήθειας ώστε να προβλέπονται περισσότερες ευκαιρίες για τις γυναίκες οικονομικά να ενεργοποιηθούν και ταυτόχρονα υλοποιούμε και την ανάλυση αντικτύπου στην οικονομία από την ισότητα γιατί οποιαδήποτε νομοθεσία θα περάσει από τη Βουλή μας περνάει από αυτή την ανάλυση για να έχουμε μια συνολική εικόνα. Η Βουλή είναι βεβαία και απεπισμένη ότι αυτοί οι νόμοι πρέπει να περάσουν για να καταγράφουν σωστά τις διαφορές που αντιμετωπίζουν στην ζωή τους επαγγελματικοί και καθημερινοί άντρες και γυναίκες. Δεν μπορεί να είμαστε ε, κοφή προς τις πραγματικές ανάγκες των ανθρώπων στην νομοθεσία. Επίσης, επικεντρώνουμε την προσοχή μας στην καταπολέμηση αυτού του μισθολογικού χάσματος με τη δημιουργία των κατάλληλων μηχανισμών για να υπολογίσουμε και να αναλύσουμε πόσο είναι αυτό, πόσο μεγάλο είναι, σε ποιους τομείς εντοπίζεται κυρίως πώς μπορούμε να χτυπήσουμε το κακό στη ρίζα του τη σωστή στιγμή και πώς μπορούμε να έχουμε τη σωστή ανάλυση για να ξέρουμε τι να το κάνουμε για να το χτυπήσουμε. Μια άλλη σημαντική πρωτοβουλία που αναλάβαμε πρόσφατα είναι η καταρτισμό του προπολογισμού βάσει του φύλου. Ο έμφυλος προϋπολογισμός. Ε, είναι ένα προηγμένο στάδιο ε, της δουλειάς μας. Κάνουμε ό,τι μπορούμε, αλλά αυτό που έκανε η Βουλή, αυτό που έκανε το Κοινοβούλιο μας, είναι ότι εφήβρε μια πολύ καλή μεθοδολογία που είναι ένα χρησιμότατο εργαλείο ώστε η εκτελεστική εξουσία να εντοπίσει ποια προγράμματα εντός του προπολογισμού έχουν ιδιαίτερη σκοπιμότητα, ιδιαίτερη σημασία μάλλον για τη διάσταση του φύλου και εκεί τους δίνει ένα, μια ενίσχυση, ένα σπρόξιμο για να μπορέσουν τα προγράμματα αυτά με ιδιαίτερη σημασία για τη διάσταση του φύλου να λειτουργήσουν καλύτερα. Το πιλωτικό του στάδιο, το πιλωτικό του τρέξιμο θα μας επιτρέψει να πονήσουμε καλύτερους προπολογισμού που λαμβάνουν υπόψη τη διάσταση του φύλου. η εκτέλεση, ο σωστό σχεδιασμό και η εκτέλεση ενό τέτοιου προπολογισμού θα επιτρέψει να ενισχυθεί ισότητα το φύλου γενικώ όλη τη χώρα. Το τελευταίο, αλλά όχι λιγότερο σημαντικό, το ανέφερα και στην αρχή, ήθελα να σα πω δύο λόγια για τη θεσμική διάσταση. Τι φορεί εργάζονται για να φέρουν ει όλα αυτά που έχουμε να κάνουμε, που είναι πολλά. Έχουμε δύο βασικού μηχανισμού στο επίπεδο του Κοινοβουλίου και του, της κυβέρνησης. Το Συμβούλιο της Ισοσύντας των Φύλων στη Βουλή μας νομοθετεί, ελέγχει, καλεί την κυβέρνηση να λογοδοτήσει, αναπτύσσει τις βασικές πολιτικές κατευθύνσεις για την ισότητα των φύλων. Όμως έχουμε και έναν εξαιρετικό μηχανισμό στο επίπεδο της εκτελεστικής εξουσίας. Την, δια, ε, την οριζόντια μάλλον υπηρεσία ελέγχου η οποία κοιτάζει τι γίνεται σε όλα τα υπουργεία και τι υπηρεσίε για να δει κατά πόσο εφαρμόζεται η πολιτική που έχει εγκρίνει το Κοινοβούλιο. Και το τρίτο επίπεδο που προσπαθούμε να αναπτύξουμε τώρα κιόλα είναι τα τοπικά συμβούλια σε επίπεδο αρχών τοπική αυτοδιοίκηση. Σε επίπεδο κοινοτήτων, δήμων και πόλεων. Έχουν διαφορετικό ρόλο μεν, αλλά είναι πολύ σημαντικά. Διότι τα συμβούλια αυτά είναι πολύ πιο κοντά την ε, τοπική πραγματικότητα, στη ζωή των πολιτών. Καταλαβαίνουν τις ανάγκες και ε, τις ελλείψεις σε πολύ καλύτερο βαθμό από ό,τι εμείς και μπορούν να διαμεσολαβήσουν για να αντιμετωπιστούν οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στο τοπικό επίπεδο, στην πράξη. Το Συμβούλιο Εσότητα των Φίλων, τα, τα Συμβούλια τα Δημοτικά, είναι καλύτερα σε θέση να ε, μελετήσουν τα προβλήματα αυτά, να τα προβάλλουν σωστά και να ε, λάβουν μέτρα. Τα προγράμματα αυτά έχουν στηριχθεί από το Ευρωκοινοβούλιο. Έχει υποστηριχθεί οριζόντια ομάδα δράση σε λειτουργικό, λειτουργικό επιχειρησιακό επίπεδο. Ε, τους, έχει ενθαρρύνει πολύ του διάφορου φορεί να κάνουν αποτελεσματικά τη δουλειά του ώστε τα αποτελέσματά μας να είναι, καρποφο... να είναι καλά και συστηματικά σε καθημερινό επίπεδο. Μας έχει βοηθήσει πολύ με το ε, Κοινοβουλευτικό Συμβούλιο για την Ισότητα των Φύλων, με την καταπολέμηση της έμφυλης βίας, με την έγκριση αυτού του σημαντικότατου νομοσχεδίου για ε, το νόμο κατά τη διακριτική μεταχείριση και τη σχολική παρενόχληση των γυναικών και για τις πολύ σημαντικές εκστρατείες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης που έχουμε οργανώσει. Ήταν κέρια σημασία όλα αυτά για να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα προβλήματα στη χώρα μας. Τη χαμηλή πολιτική συμμετοχή, την εμφυλιβία, τη σεξουαλική παρενόχληση. Μέχρι προσφάτως ήταν κάτι που ο κόσμος δεν το παραδεχόταν καν ότι υπάρχει. Δεν το βλέπω ως πρόβλημα. και εκστρατείε για την ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση, τα προγράμματα που υποστηρίζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ζωτική σημασία για όλα τα αποτελέσματα που επιτύχαμε και για όλη μας τη δουλειά. Έχουμε μια κοινωνία πολύ εύρωστη και πολύ δυναμική. Ε, ο ρόλος της εδώ είναι καθοριστικός. Αλλά και η, Ένωση, η Ευρωπαϊκή Ένωση του στήριξε όχι μόνο στους κρατικούς φορείς δηλαδή, αλλά και στις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών. Αυτό είναι ένας φανταστικός συνδυασμός για να καταφέρουμε όσα καταφέραμε. Μια καλή επικόνηση για το πόσο καλά τα έχουμε πάει και πόσο πρόοδο, πόση πρόοδο έχουμε επιτελέσει. Είναι ότι πριν από μερικά χρόνια το να χρησιμοποιεί κανείς τον όρο φίλο ήταν κακό. Ξύνιζαν τα μούτρα τους όταν άκουγαν να λέει κανείς gender, φίλο. Η γάμη μεταξύ ανηλίκων. Η απαγωγή για να παντρέψουν τα κορίτσια. Το θεωρούσαν κάτι κανονικό, φυσιολογικό. Τώρα, για τις γυναίκες της Γεωργίας, για όλους δηλαδή στη Γεωργία, θεωρείται ποινικό αδίκημα. Ούτε που θα παίρνει από το μυαλό κανένα να κάνει κάτι τέτοιο. Και τα νεαρά κορίτσια θέλουν να είναι φεμινίστριες. Θέλουν να εργαστούν για τα δικαιώματα των γυναικών, για τις υποθέσεις και τα πράγματα των γυναικών. Αυτό για μένα είναι η καλύτερη απόδειξη ότι έχουμε προχωρήσει. Τα κορίτσια ήταν... Τα κορίτσια που πίστευαν ότι ο γάμος ε, πρόωρη είναι το καλύτερο που του συμβεί, τώρα θέλουν να εργαστούν, θέλουν να βρουν δουλειά, θέλουν ε, να έχουν δικαιώματα, να είναι ισχυρέ και ανεξάρτητες. Αυτό το πετύχαμε και χάρη στη δική σα στήριξη. Το εκτιμούμε πολύ και σας ζητούμε να ε, παρακολουθείτε την πρόοδο αυτή και να συνεχίσουμε την αγαστή συνεργασία που είχαμε στην παράδο των ετών. Σα ευχαριστώ πολύ και στη διάθεσή σα για απαντήσει. Mm, σα ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω τώρα το λόγο στα μέλη. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ε, Σας ευχαριστώ λοιπόν ε, πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, χαίρομαι πολύ που λαμβάνει σήμερα αυτή η ακρόαση χώρα έτσι ώστε να έχουμε τη δυνατότητα να ακούσουμε τους ε, συναδέλφους από τη Γεωργία προκειμένου να ακούσουμε πώς διαμορφώνεται η πολιτική ε, των φίλων εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα ήθελα να σας ε, συγχαρώ γιατί όλα αυτά που μας διηγηθήκατε μόλις ε, τώρα μας κάνουν μεγάλη εντύπωση. Ήθελα να σας ρωτήσω πώς θα καταφέρατε ε, να φτάσετε σε ένα τόσο καλό αποτέλεσμα. Γιατί αν σας άκουσα καλά, αυτή η δομή αν των διαφορετικών θεσμικών οργάνων η οποία ε, επιλαμβάνεται ακριβώ των ζητημάτων ισότητα του φύλου στο κοινοβούλιο σας, στις διάφορους ε, οργανισμούς τοπικής και περιφερειακής ε, αυτοδιοίκησης είναι ένα πραγματικό επίτευγμα. Είναι κάτι δηλαδή το οποίο θέλουμε και εμεί να επιτύχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και δεν το καταφέρνουν όλα τα κράτη-μέλη. Δεν έχουν δηλαδή ένα τέτοιο δίκτυο θεσμικών οργάνων και γενικότερα οντοτήτων. Ε, πραγματικά δηλαδή πρόκειται για μια ε, τεράστια επιτυχία αυτή την οποία μας διηγηθήκατε. Άρα λοιπόν αυτή η ε, ειδικότερα πολιτική καταπολέμηση της εισβίας και το γεγονός ότι τονίζεται ιδιαίτερα είναι κάτι το πολύ σημαντικό. Επίσης είναι πολύ θετικό το ότι πράγματι κινείστε πάντοτε προς την ισόρροπη εξορρόπηση των δύο φύλων. Δηλαδή, εάν θέλουμε να επιτύχουμε κάτι, ε, τότε πρέπει να ξεκινήσουμε πάντοτε από εκεί να ξεκινάμε. Δηλαδή, από την καταπολέμηση της βίας ε, εις βάρος των γυναικών. Γιατί δεν μπορεί να υπάρξει κανένας ο οποίος ε, δημοσίως θα ταχθεί κατά μέτρων αυτή τη φύση, δηλαδή για την καταπολέμηση τη βία εις βάρος των γυναικών. Είναι λοιπόν θετικό το γεγονό ότι η Γεωργία τα κάνει όλα αυτά, το γεγονό ότι έχει κυρώσει και τη σύμβαση της Κωνσταντινούπολη γιατί και αυτό είναι πολύ σημαντικό και σας συγχαίρω για αυτή την ε, κύρωση δηλαδή της ε, σύμβουσης καθώς ε, έλαβε χώρα σχετικά αργά. Θα ήθελα να σας ερωτήσω σε αυτό το πλαίσιο εάν καταφέρατε να πείσετε κάποιους από τους πιο επιφανείς πολιτικούς άντρες ε, της Γεωργίας να προσυπογράψουν τέτοιου είδους πολιτικές για την ισότητα των φίλων. Γιατί βέβαια συνήθως ε, έχουμε να κάνουμε με άντρες οι οποίοι τελικά λαμβάνουν αυτές τις ε, αποφάσεις. Οπότε είναι σημαντικό να συγκεντρώσουμε και από την τους πλευρά υποστήριξη. Οπότε θα ήθελα πολύ να μάθω κατά πόσο η δουλειά που κάνατε εσείς από την πλευρά, αν θέλετε, των γυναικών, ε, έχετε καταφέρει να ενταχθεί ε, στις, στις βασικές πολιτικές της γεωργίας ε, και σε όλους εκείνους δηλαδή τους τομείς όπου οι υψηλότερες θέσεις καταλαμβάνονται από άνδρες. Θα πρέπει δηλαδή σε αυτό το πλαίσιο όλες οι διαφορετικές πολιτικές που λαμβάνουν ε, υπόψη το ε, φύλλο να εφαρμόζονται με τον σωστό τρόπο. Η κυρία Μούντι έχει τώρα το λόγο. Σας ευχαριστώ ε, πολύ και σας ε, καλωσορίζω εδώ στην ε, Επιτροπή ΙΦΕΜ. Χαίρομαι πολύ που είστε εδώ. Και θα ήθελα να αναφερθώ στα όσα αναφέρατε στην ομιλία σας. Καταρχήν να αναφερθήκατε λίγο εδώ στο ιστορικό. Και με βάση την ιστορία σας να σας πούμε ότι υπήρχε ε, καθολικό δικαίωμα ε, ψήφου, δηλαδή και για τις γυναίκες και για τους άντρες, ε, τα καταφέρατε εσείς πιο πριν από εμάς. Εμείς δηλαδή ξεκινήσαμε από το 20 και μετά, οπότε πραγματικά το, τα καταφέρατε νωρίτερα από εμάς. Από εκεί και μετά, εγώ γνωρίζω πως η πρόεδρος που εξελέγει στην Γεωργία ε, είναι όχι μόνο γυναίκα, αλλά και μουσουλμάνα. Οπότε πραγματικά θα πρέπει εδώ να σας ε, ε, συγχαρούμε για όλα αυτά, σε ό,τι αφορά την ιστορία σας. Τώρα, εγώ είμαι κάπως εξοικειωμένη με τη γεωργία και εκείνο που με εκπλήσει πάντοτε είναι η ποιότητα και η ισχύ των ε, γυναικών ε, της Γεωργίας. Και αυτό το διαπιστώνω βέβαια και ε, στο κοινοβούλιο σας, αλλά και στην κοινωνία των πολιτών. Βλέπουμε δηλαδή εκεί που υπάρχουν πολλές χειρές γυναίκες. Επίσης έχετε πρόεδρο, γυναίκα όπως είπατε, και μόνο το 8% των αρχικών κρατών και κυβερνήσεων ανά τον κόσμο είναι γυναίκες. Οπότε και αυτό σας διακρίνει. Επίσης και η πρέσβυρά σας εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ε, γυναίκα και πολύ εντυπωσιακή και εκείνη. Οπότε πραγματικά από τη δική σας πλευρά καταδεικνύεται ε, την αξία του να υποστηρίζουμε τις γυναίκες. Και το πόσο θα πρέπει να καταλαμβάνουν ε, τέτοιες σημαντικές θέσεις, σημαντικά πόστα στη Γεωργία. Επίσης σα συγχαίρω για τη δουλειά που έχετε κάνει σε ό,τι αφορά την καταπολέμηση της βία ει βάρο των γυναικών, γιατί αυτό που έχει καταδείξει η επιτυχία αυτού του, του project, αν θέλετε, από τη δική σας πλευρά, είναι η επιβολή της νομοθεσίας και η κατάλληλη, δηλαδή, εποπτεία σε ό,τι αφορά την επιβολή της νομοθεσίας. Και νομίζω πως θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμο για όλους μας να τονιστεί αυτό, δηλαδή το πώς η, συγκεκριμένη ενότητα, η μονάδα που δημιουργήθηκε μέσα στο Υπουργείο Δικαιοσύνη ε, έπαιξε το σημαντικό ρόλο σε ό,τι αφορά την επιβολή αυτή τη νομοθεσία για την καταπολέμηση τη βία κατά των γυναικών. Επίση, αναφερθήκατε ε, στο ζήτημα ε, των διακρίσεων και τη σεξουαλική επαρενόχληση και των νομοσχεδίων που έχουν υποβληθεί. Θα ήθελα να μα ενημερώσετε λίγο παραπάνω προ το τι ακριβώ συμβαίνει, ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα πότε προβλέπετε ότι θα υπάρξει εφαρμογή αυτής της νομοθεσίας. Και εδώ ε, βέβαια ε, τονίζω ότι υπάρχει πραγματική συμμετοχή και της ε, κοινωνία των πολιτών. Ε, τώρα, σε ό,τι αφορά την πολιτική δράση, αν θέλετε, τη συμμετοχή των, στην πολιτική ζωή των γυναικών. Πράγματι έχετε γυναίκα πρόεδρο, από την άλλη πλευρά όμως στις δημοτικές εκλογές της Περσινές δεν είχατε πολλές γυναίκες οι οποίες εξελέγησαν και ποιοι άλλοι τρόποι μπορούν να ε, υπάρξουν από τη δική μας πλευρά προκειμένου να προωθηθεί νομοθεσία προς αυτή την κατεύθυνση. Γιατί γνωρίζετε πόσο και γνωρίζουμε πολλοί από τις ε, χώρες μας πόσο σημαντικό είναι να υπάρχουν ποσοστώσεις σε ό,τι αφορά την εκπροσώπηση των γυναικών. Και τέλος, γιατί νομίζω ότι μακρηγόρησα, σε ό,τι αφορά την απόδοση αυτοεξουσιότητα, αυτό το empowerment στι γυναίκε σε οικονομικό επίπεδο. Νομίζω πως ε, τα τοπικά συμβούλια για το φύλλο θα παίξουν έναν καθοριστικό ρόλο, γιατί ακριβώς θα αναλαμβάνουν δράσεις σε τοπικό επίπεδο και σε εκείνο το τοπικό επίπεδο θα επιτύχετε το ταχύτερο αντίκτυπο, αν όχι και το μεγαλύτερο. Οπότε, Σα ρωτώ, μπορούμε να κάνουμε περισσότερα από την πλευρά τη Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να σας υποστηρίξουμε. Και σε ό,τι αφορά επίσης την νομοθεσία, σε ό,τι αφορά την ισότητα των μισθών μεταξύ των δύο φύλων. Έχουν υπάρξει μια σειρά από αποφάσεις ε, του ε, Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ό,τι αφορά ακριβώς ε, την ίδια αμοιβή ε, για την ίδια εργασία, για τον, την ίδια αξία εργασίας ε, και ό,τι καθεξής. Ε, αυτά από την πλευρά μου και σας ευχαριστούμε πολύ που είσαστε σήμερα εδώ και παρουσιάσατε την σημαντική δουλειά που κάνετε και που την παρουσιάσατε σε εμά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. Δίνω τώρα το λόγο στην κυρία Τζουλουγούρ. Σας ευχαριστώ πολύ. Πραγματικά ήταν καταπληκτικά τα όσα μας αναφέρατε και μας υπενθυμίζουν νομίζω πως ε, ε, Ορισμένε φορές δεν είναι καλό να είμαστε έτσι ευρωκεντρικοί, να εστιάζουμε μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς υπάρχουν και πολύ χρήσιμα παραδείγματα από τα όσα συμβαίνουν εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης Και από εκείνα τα παραδείγματα μπορούμε και εμεί να αντλήσουμε κάποια διδάγματα για μας από άλλες χώρες. Άρα λοιπόν η παρουσία σας σήμερα εδώ μας βοηθάει να αναλογιστούμε λίγο το πώς μπορούμε να είμαστε καλύτεροι στα όσα κάνουμε σε αυτό το τομέα. Εγώ σκεφτόμουν λίγο τη γεωγραφική θέση της γεωργίας και αναλογιζόμουν το πόσο μεγάλη επίδραση μπορείτε να έχετε στις χώρες ε, της γειτονικές σας, της ευρύτερης ε, περιοχής όπου έχουμε πολύ σας, αν θέλετε ε, αρχηγούς κρατών και οι οποίοι κάνουν κάποια πολύ αποκρουστικά πράγματα σε ό,τι αφορά την ισότητα των φύλων, αλλά και σε ό,τι αφορά τη διαφάνεια, σε ό,τι αφορά τη δημοκρατία και ούτω καθεξής. Οπότε, όταν βλέπουμε να μεταβάλλεται η παγκόσμια τάξη ε, και εγώ μόλις ε, τώρα προσήλθα εδώ από μια διάσκεψη που είδαμε σε ό,τι αφορά την απονόμηση των δικαιωμάτων, την απονόμηση των, των γυναικών αλλά και των ΛΟΑΔΜΕ και ούτω καθεξής ε, και την αύξηση εδώ του εθνικισμού, τα ζητήματα σε ό,τι αφορά την κλιματική αλλαγή. Διαπιστώνω λοιπόν ε, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση συχνά αναφέρεται στην χριστιανοδιδαϊκή ε, προέλευσή της αν θέλετε, αλλά δεν λαμβάνει υπόψη της άλλα παραδείγματα, άλλες υπέροες, πράγμα το οποίο θεωρώ πως είναι πολύ επικίνδυνο ως στάση την οποία έθετε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν λοιπόν ακούω τα όσα συμβαίνουν στη Γεωργία, τα όσα εντυπωσιακά κάνετε και λαμβάνοντα υπόψη τι προκλήσει που αντιμετωπίζουν οι χώρε εκείνη τη ε, περιοχή, ε, θα ήθελα να μα πείτε λίγο πώ σκοπεύετε να, ε, να αναλάβετε έναν ηγετικό ρόλο εδώ, αν θέλετε. Ε, κάτι το οποίο χρειαζόμαστε δηλαδή και εμείς εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ έχω εργαστεί πολύ στην Ουκρανία και γνωρίζω πως υπάρχουν πολλοί καλοί άνθρωποι στην Ουκρανία οι οποίοι προσπαθούν να αλλάξουν τα πράγματα εκεί. Δηλαδή οι γυναίκες τις οποίες έχω συναντήσει στην Ουκρανία είναι καταπληκτικές, ε, έχουν, δίνουν πραγματικό αγώνα. Ε, και το λέω αυτό βασιζόμενοι σε, σε διαφορετικούς λόγους και ε, συμμετέχω από την πλευρά ε, τη δική μου ως Ευρωβουλευτής και για τα δικαιώματα των ΛΟΑΔΜ και είχαμε κάνει μια πολύ ενδιαφέρουσα συνάντηση με βουλευτές ε, της Ουκρανίας προκειμένου να προσπαθήσουμε να ενθαρρύνουμε τους βουλευτές αλλά και τους υποψήφιους ε, βουλευτές της Ουκρανίας να αντιληφθούν καλύτερα τα ανθρώπινα δικαιώματα και συγκεκριμένα τα δικαιώματα των ΛΟΑΔΜ. Οπότε δεν ξέρω αν έχετε κάποια σχέση εκεί με την ελόγω οργάνωση ε, της Ουκρανίας, αλλά θεωρώ πως είναι μια πολύ καλή οργάνωση, ε, καθώς ε, μέσω αυτής μπορούν να συνεργαστούν βουλευτές από όλο τον κόσμο σε ό,τι αφορά τα ζητήματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας. Ευχαριστούμε, Τζούλη Word. Τώρα, συνεχίζουμε. Η κυρία Σουκασλίδη θα πρέπει να λάβει τις ευχαριστίες μας που μας έδωσε την ευκαιρία να κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Όσον αφορά την ισότητα των δύο φίλων, η Γεωργία έχει κάνει πολλά πράγματα. Το ξέρω, γιατί εγώ είμαι από τη Λιθουανία. Και η σχέση ανάμεσα στη Λιθουανία και την Γεωργία είναι σχέσεις που ήταν πάντα ιδιαίτερα ισχυρε και φιλικές. Είμαστε φίλες χώρες και στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ισότητας των δύο φίλων, της οικονομικής, πολιτιστικής συνεργασίας. Οι σχέσεις μας πάντα ήταν ισχυρές και στενές. Οπότε σας καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά. Καταλαβαίνω πολύ καλά αυτό που λέτε, ότι δηλαδή ε, τι ευφυΐα χρειάζεται για να αλλάξουμε τα πράγματα, για να γίνει δεκτό ότι οι γυναίκες είναι ίσες με τους άντρες και ότι μπορούν εξίσου να συμμετέχουν στην πολιτική, την οικονομική, την κοινωνική ζωή. Οπότε εγώ είμαι πολύ περήφανη για σας. Είμαι περήφανη γιατί η Γεωργία έχει κυρώσει τη σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, ενώ υπάρχουν χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν το έχουν κάνει αυτό ακόμα. Εσείς λοιπόν μπορείτε να αποτελέσετε ένα καλό παράδειγμα για άλλες χώρες, ακόμα και για χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εσείς θα έχετε ε, κοινοβουλευτικές εκλογές του χρόνου, έτσι. Και είπατε ότι από τους βουλευτές οι γυναίκες είναι το 15% στη Βουλή σας. Ε, εύχομαι στο νέο κοινοβούλιο να είναι πολύ περισσότερες. Την επόμενη εβδομάδα λοιπόν εμείς θα γιορτάσουμε την ημέρα της γυναίκας. Εκείνη την ημέρα λοιπόν, εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θα συζητήσουμε για το τι αποφάσεις πρέπει να υιοθετήσουμε μαζί, ώστε να έχουμε περισσότερες γυναίκες στην πολιτική ζωή, εδώ, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στα εθνικά, στα τοπικά κοινοβούλια είναι ο μόνος δρόμος που μπορεί να μας βοηθήσει να πάρουμε τις αποφάσεις εκείνες οι οποίες θα οδηγήσουν στην ισότητα μεταξύ των δύο φύλων. Θέλω να σας ρωτήσω, λοιπόν, τι γίνεται με την απασχολησιμότητα των γυναικών, τη δυνατότητα απασχόλησης, δηλαδή βρίσκουν εύκολα δουλειά οι γυναίκες, έχουν την δυνατότητα να συνδυάσουν ε, την ιδιωτική τους ζωή με την επαγγελματική, τη σταδιοδρομία τους, δηλαδή με την οικογένειά τους. Επίσης, θέλω να σας ρωτήσω πώς βλέπετε την δική μας μελλοντική συνεργασία Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δηλαδή και Κοινοβουλίου της Γεωργίας, για να ανταλλάσσουμε βέλτιστες πρακτικές. Αυτά από τη δικιά μου την πλευρά. Άλλος κανείς έχει ερωτήσει, σχόλια. Λοιπόν, έχετε πέντε λεπτά για να απαντήσετε σε ερωτήσεις μας. Σας ακούμε. Σας ευχαριστώ πολύ πραγματικά για τα ενθαρρυντικά σας λόγια. Πραγματικά τα χρειαζόμαστε, τα χρειάζεται κανείς κάθε τόσο, γιατί η δουλειά που κάνουμε έχει δυσκολίες. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, με ρωτήσατε για την κύρωση της σύμβασης της Κωνσταντινούπολης. Η κύρωση έγινε το 2017 αλλά ε, πήρε δύο χρόνια στο Υπουργείο Δικαιοσύνης ώστε να καταλήξουμε σε μια αλλαγή προπτικής. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι πρέπει να προχωρήσουν τα πράγματα, όχι μόνο ώστε επίσημα ε, να γίνεται η κύρωση, αλλά να υλοποιείται και όλα το περιεχόμενο της σύμβασης. Η υλοποίηση λοιπόν, η εφαρμογή είναι το στοιχείο κλειδί. Το πιο σημαντικό κομμάτι όλες τις διαδικασία γιατί μπορεί να έχουμε στο χαρτί διάφορα, αλλά δεν σημαίνει ότι έχουμε και αποτελέσματα. Οπότε το εργαλείο αυτό εφαρμογής, το ότι περάσαμε τόσο χρόνο προσπαθώντας να σκεφτούμε πώς θα εφαρμοστεί καλύτερα το περιεχόμενο της σύμβασης, αυτό ήταν το φοβερό. Και συνεισέφεραν πολλοί συνάδελφοι σε αυτό. Η αλήθεια είναι ότι είμαστε τυχεροί δεν έχουμε ε, πολλούς, αλλά σίγουρα έχουμε αρκετούς αφοσιωμένους άντρες συναδέρφους που μας βοηθούν πολύ. Το θέμα της ισότητας ε, των ε, φίλων, η σχετική επιτροπή αποτελείται από 17 μέλη και μόνο τρεις είναι άντρες. Μας βοηθούν όμως πολύ κάθε φορά που τους χρειαζόμαστε. Για παράδειγμα, για να περάσει νομοθεσία για τη σεξουαλική όχληση. Όπως επίσης και η τροποποίηση της ε, νομοθεσίας για τη μη διάκριση. Συμφωνούμε λοιπόν έτσι με τους συναδέρφους μας τους άντρες ότι και αυτοί πρέπει να πιέσουν υπέρ της νομοθεσίας ή εκείνοι πρέπει να αναλάβουν κάποια πρωτοβουλία, εκείνοι να παρουσιάζουν στις επιτροπές τις πρωτοβουλίες αυτές και να φροντίζουν να φτάσουν στην Ολομέλεια. Μέχρι τώρα λειτουργήσε. Και αυτή η νομοθετική πράξη που προτάθηκε από τους άντρες οδηγεί σε μεγαλύτερη ακόμα αποδοχή από ότι αν η πρόταση είχε έρθει από γυναίκες, από φεμινίστριες. Μέχρι τώρα λοιπόν λειτουργήσε αυτή η μέθοδος και μας έχει στηρίξει και η Προεδρία του Κοινοβουλίου, έγινε σχετική δήλωση και σίγουρα πρωταγωνιστούν οι γυναίκες με κάποιες εξαιρέσεις που φυσικά και είναι ιδιαίτερα λαμπρές και σημαντικές για μας και μακάρι να γινόταν πιο συχνά. Για την ερώτηση της Κλέρ τώρα, για τις υποχρεωτικές ποσοστώσεις και για την σεξουαλική όχληση. Σας ξεκινήσω από αυτό. Εμείς έχουμε ακροάσει στην Επιτροπή μας και σύντομα θα φτάσει το θέμα και στην Ολομέλεια. Μόλις ξεκίνησε η διαδικασία, πριν από λίγες εβδομάδες, και ελάχιστο χρόνος για να περάσει η νομοθεσία είναι περίπου τρεις μήνες. Που σημαίνει ότι έχουμε αυτό το διάστημα μπροστά μας, δηλαδή σε τρεις-τέσσερις μήνες θα περάσει η νομοθεσία και εφόσον έχει περάσει υπάρχει ο μηχανισμός εφαρμογής γιατί προβλέπονται τέτοιοι μηχανισμοί από το Υπουργείο Εσωτερικών και τον Ομπουτσμαν. Ε, Οπότε οι μηχανισμοί υπάρχουν. Μετά από τρεις-τέσσερις μήνες που θα περάσει θα αρχίσει η κυλοποίηση. Όσον αφορά τώρα τις ποσοστώσεις πρέπει να τις εισάγουμε στον νόμο. Χρειαζόμαστε να επαναδιατυπωθεί το σχέδιο, γιατί απέτυχε την πρώτη φορά, και να επαναπροταθεί στο Κοινοβούλιο. Βέβαια δεν μπορούμε συγχρόνως να περάσουμε όλα σε αυτές τις νομοθετικές πράξεις, γιατί είναι πολύ για τους βουλευτές μας. Οπότε προσπαθούμε να προχωρήσουμε βήμα-βήμα. Θα αρχίσουμε τη διαδικασία όσο γίνεται πιο γρήγορα εφόσον έχουμε τελειώσει με τη σεξουαλική όχληση. Μόλις περάσει αυτή η νομοθεσία, τότε θα ξεκινήσουμε με τις υποχρεωτικές ποσοστώσεις για την ισότητα μεταξύ των δύο φύλων. Μέχρι τώρα η μέθοδος αυτή έχει αποφέρει καρπούς. Οι βουλευτές έτσι μπορούν να στηρίξουν τις πρωτοβουλίες μας τώρα όσον αφορά ε, τις οικονομικές επιπτώσεις της, ε, των γυναικών που βρίσκονται σε διευθυντικές θέσεις. Βάζουμε ως προτεραιότητα διάφορα θέματα. Επαγγελματική κατάρτιση, πρώτα απ' όλα, είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και είναι κάτι το οποίο έχει λειτουργήσει υπέρ της απασχόλησης των γυναικών η επαγγελματική κατάρτιση. Αναλύουμε λοιπόν τώρα ποια είναι τα προγράμματα που θα έπρεπε να επαναλάβουμε, να αυξήσουμε και πού στη χώρα. Και τώρα προσπαθούμε να δούμε διάφορα κρατικά προγράμματα, πώς έχουν συνεισφέρει στην ε, οικονομική ενίσχυση των γυναικών και πόσο βοηθούν τις γυναίκες που τα θέλουν. Οι στατιστικές απασχόλησης η πρόεδρος με ρώτησε γι' αυτό, δείχνουν ότι 58% των γυναικών είναι οικονομικά δραστήριες, ενώ στους άντρες το ποσοστό αυτό είναι 75%. 42% των γυναικών είναι αδρανείς οικονομικά, ενώ μόνο 25% των ανδρών είναι σε αυτή την κατηγορία. Τα τελευταία χρόνια είχαμε μεγαλύτερη αύξηση στις γυναίκες που δραστηριοποιούνται οικονομικά από ό,τι στους άντρες αλλά η διαφορά των ε, μισθών είναι περίπου στο 40%. Δεν είναι ακριβές βέβαια αυτό το νούμερο. Κάθε μισθός γυναικών είναι περίπου 700-800, ενώ για τους άντρες είναι 1000-1100. Οι διαφορές λοιπόν είναι μεγάλες. Και αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να μειώσουμε αυτό το χάσμα το πρώτο που πρέπει να κάνουμε είναι να έχουμε ε, στοιχεία, δεδομένα, ε, στατιστικά δεδομένα, ακριβή, για να μπορούμε να εντοπίσουμε με ακρίβεια το φαινόμενο. Όσον αφορά τις γείτονες χώρες, η Γεωργία ξέρει ξεκάθαρα που θέλει να βρεθεί και θέλει να βρεθεί μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό είναι που μας βοηθάει να προχωρήσουμε και χαιρόμαστε πολύ να μοιραζόμαστε τις εμπειρίες μας ε, με τους γειτονές μας. Αλλά οι γειτονικέ χώρες, οι πολιτικές ε, σίγουρα επηρεάζουν πολύ, αλλά ελπίζουμε η Γεωργία να καταφέρει να αποτελέσει ένα θετικό παράδειγμα, γιατί έχει πραγματικά καταπληκτικές γυναίκες, κοινωνία των πολιτών, οι μη κυβερνητικές ε, οργανώσεις, γυναίκες, τα κορίτσια στη Γεωργία είναι πιο ομορφωμένα σήμερα. Έχουν μελετήσει, ενημερώνονται. Δυστυχώς όμως καταλήγουν να είναι ανενεργά οικονομικά. Παρόλο που την, την περισσότερη δουλειά την κάνουν οι γυναίκες, τις αποφάσεις τις παίρνουν οι άντρες. Ε, αυτό πρέπει να αλλάξει. Και κάθε φορά, σε κάθε εκλογέ, τοπικέ εθνικέ θέλουμε να δημιουργήσουμε την αναγκαία ισορροπία. Πρέπει να υπάρχει προκειμένου να προδεύσει πιο γρήγορα η χώρα μας. Νομίζω ότι λίγο πολύ έχω απαντήσει στις ερωτήσεις σας. Για άλλη μια φορά θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την ευκαιρία που μου δώσατε, για τη στήριξή σας και το έτοιμά μου είναι και πάλι να συνεχίσουμε αυτή την τόσο καλή συνεργασία που έχουμε με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Διότι κάνει πραγματικά τη διαφορά, την κάνει για μας και αξίζει τον κόπο να επενδύσει κανείς αυτή την ενέργεια, αυτή την προσπάθεια γιατί έτσι αλλάζει η χώρα. Έτσι αλλάζει η ζωή των ανθρώπων. Πολύ σημαντικό αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ λοιπόν που μου δώσατε την ευκαιρία αυτή σήμερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσίασή σας όσον αφορά την κατάσταση στην ε, Γεωργία. Όντω έχουμε πολύ καλή συνεργασία μεταξύ μας.

Πρόεδρος, ε, συνεχίζουμε με την συνεδρίασή μας. Το επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη, το σήμερα 5, είναι 50, 50 ε, εκστρατεία ε, τα λόμπι Ευρωπαίων γυναικών. Το λόμπι αυτό θέλει τη συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θέσεις υψηλού επίπεδου για τις γυναίκες στην απασχόληση. Θα δώσω το λόγο στην κυρία Γκνέβεν Λεβαμπρέντ, η οποία είναι πρόεδρος του λόμπι αυτού. Έχετε 10 λεπτά στη διάθεσή σας. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Καταρχήν, κυρία Πρόεδρε της Επιτροπής ΦΕΜ, θα ήθελα να σε ευχαριστήσω για τη δυνατότητα που μας δίνετε να παρουσιάσουμε εδώ την εξταθιά μας. Λέγομαι Κβεντολίνο Εφεύ και έχω εκλεγεί ως ε, πρόεδρος ε, της EWA ε, από τον περσινό Ιουνιό και όπως ίσως θα γνωρίζετε αυτό το λόμπι είναι η μεγαλύτερη γενική οργάνωση για την δικαιώματα των γυναικών που προωθεί ακριβώς την ισότιμη μεταχείριση και τα ίσα δικαιώματα για τις γυναίκες και τους άντρες και μέλη εδώ μπορούν να είναι ε, να προέρχονται από, όλες ε, τις, από όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υποψήφιες σε χώρες προς προσχώρηση. Και έχουμε 28 εμ, οργανώσεις ε, παγκόσμιες οι οποίες συμμετέχουν, ενώ εκπροσωπούμε 2.000 συνολικά οργανώσεις για την προστασία των δικαιωμάτων των γυναικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, κυρία Πρόεδρε, τον περασμένο μήνα βρεθήκαμε στη δική σας πατρίδα, όπου ρωτήσαμε τα μέλη μας ως προς το πώς έχει η κατάσταση στις διάφορες ε, χώρες ε, ε, σε σχέση με τις γυναίκες και τα δικαιώματα των γυναικών. Και σχεδόν όλοι μας είπαν ότι εδώ υπάρχει πολιτική ατζέντα, πολιτικές προτεραιότητες τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ότι εκείνος ο οποίος εκλέγεται, εκείνος ο οποίος βρίσκεται στην ηγεσία παίζει καθοριστικό ρόλο σε ό,τι αφορά ακριβώς την ε, προστασία των δικαιωμάτων των γυναικών και την ισότιμη μεταχείριση μεταξύ ανδρών και γυναικών. Αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη αντιμετωπίζουμε μία σειρά από ζητήματα, αλλά σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να έχουμε πάντοτε ένα πράγμα κατά νου. ο αριθμός των γυναικών που διαδηλώνουν μαζί μας πλέον στις, ε, ε, ε στους δρόμους ε, αυξάνεται όλο και περισσότερο και το κίνημα του Me είναι και αυτό πολύ σημαντικό και στη δική μας και σε χώρες. Και αυτή η αντίσταση από την πλευρά των γυναικών τώρα θα πρέπει να λάβει σάρκα και οστά ως πολιτικό μετασχηματισμός. Και γι' αυτό ακριβώς δημιουργήσαμε αυτήν την εκστρατεία της Ευρώπης για τις γυναίκες, οι γυναίκες και την Ευρώπη 50-50 και ε, έχουμε ξεκινήσει αυτή την ε, ε, διάδοση και την αιμορδική αυτή εκστρατεία σε όλες τις οργανώσεις μας, σε όλες τις διαφορετικές χώρες, αλλά αυτό δεν έρχεται μόνο του. Θα πρέπει να λάβουμε την υποστήριξη και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έτσι ώστε να θέσουμε την ισότητα μεταξύ των δύο φύλων στον πυρήνα της πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωση. Εκεί δηλαδή όπου θα έπρεπε να βρίσκεται ανέκαθεν. Για να το επιτύχουμε λοιπόν αυτό χρειαζόμαστε μια κοινή πολιτική στρατηγική. Χρειαζόμαστε επίσης μια πολιτική δομή για να υποστηρίξει την υλοποίηση της εν λόγω στρατηγικής. Τι σημαίνει αυτό συγκεκριμένα. Χρειαζόμαστε φυσικά στο πλαίσιο του επόμενου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μια ισχυρή επιτροπή ΦΕΜ. Επίσης, θα χρειαστούμε να υπάρξει ένας επίτροπος ή μια επίτροπος, το οποίο η μόνη αρμοδιότητα θα είναι τα δικαιώματα των γυναικών και η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών. Επίσης, θα χρειαστούμε υπουργικές διασκέψεις με θέμα ακριβώς την ισότητα μεταξύ των δύο ε, φίλων. Για παράδειγμα, υπουργοί αθλητισμού, οι οποίοι θα συναντιούνται δύο έως τέσσερις φορές ετησίως, επίσημα, ε, ή μάλλον οι Υπουργοί Αθλητισμού συναντιούνται τέσσερις φορέ επισήμω το χρόνο, αλλά το ίδιο δεν συμβαίνει με τους υπουργού που είναι αρμόδιοι για τα ζητήματα ε, ισότητας ισότητα μεταξύ των δύο φύλων. Γιατί δεν συμβαίνει αυτό, και επίση, βέβαια, χρειαζόμαστε τα απαραίτητα κονδύλια για να τα επιτύχουμε όλα αυτά. Τα κονδύλια είναι απαραίτητα για να κάνουν τη ε, δουλειά του όλε οι οργανώσει ε, για την ε, προστασία των δικαιωμάτων των γυναικών. Και επίση, βέβαια, θα χρειαστούμε και να υπάρχει ισόρροπη εξισορρόπηση μεταξύ των δύο φίλων στην επόμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Άρα λοιπόν υποστηρίζουμε αυτή την ενημερωστική μας εκστρατεία 50-50 και ποιοι είναι οι βασικοί στόχοι της. Καταρχήν να υπάρχουν περισσότερες γυναίκες οι οποίες θα ψηφίσουν. Το 2014 μόνο το 41% των γυναικών ε, ψήφισε. Ενώ το 45% των ανδρών ψήφισε. Οπότε πρέπει να έχουμε περισσότερες γυναίκες οι οποίες θα προσέλθουν στις κάλπες. Επίσης θα πρέπει να υπάρξουν άνθρωποι, περισσότεροι πολίτες, περισσότεροι ψηφοφόροι οι οποίοι θα ψηφίσουν υπέρ γυναικών και όχι απλώ γυναικών, γυναικών οι οποίε πραγματικά είναι ακτιβιστέ, θέλουν να προωθήσουν αυτή τη δουλειά. Εάν λοιπόν θέλουμε πραγματικά να υπάρξει συνέχεια στην δική μα εργασία, χρειαζόμαστε φεμινίστριε. Αυτό τι σημαίνει, σημαίνει ισόρροπη εκπροσώπηση των φίλων στους εκλογικούς καταλόγους των διαφορετικών κομμάτων και σημαίνει ότι θα πρέπει τα πολιτικά κόμματα να έχουν πολιτικά προγράμματα τα οποία λαμβάνουν υπόψη τα ζητήματα του φύλου και τα οποία προωθούνται και στις προεκλογικές τους εκστρατείες. Και αυτό βέβαια με στόχο του να υπάρχει ισόρροπη εξορρόπηση, ισότιμη εξορρόπηση μεταξύ των δύο φύλων τόσο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σε ό,τι αφορά τις ε, ηγετικές, τις ε, θέσεις ε, ε, στα θεσμικά όργανα της Ένωσης. Και, επίσης, οι πολιτικοί ηγέτε θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους τα δικαιώματα των γυναικών ως θεμελιώδε ζήτημα. Τι προτείνουμε λοιπόν εμείς για να πετύχουμε αυτούς τους στόχους. Έχουμε μία σειρά από εργαλεία που προτείνουμε. Καταρχήν, έχουμε μία, ένα έγγραφο εδώ, ε, μέσω του οποίου μπορούν να, στο το οποίο μπορούν να υπογράψουν και οι ευρωβουλευτές, εφόσον το επιθυμούν, που είναι μία δέσμευση εδώ, εδώ ο συνάδελφος από το EWL μπορεί να σας ε, διανύμει ένα αντίτυπο. Και πέραν αυτού, πέραν αυτής της δέσμευσης υπάρχει και μια έκκληση, ένα petition, το οποίο μπορούν να υπογράψουν ε, οποιοδήποτε πολίτες ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, προτείνουμε στα μέλη μας ένα kit για την άσκηση ακριβώς αυτού του lobbying, Και βέβαια μπορεί κανείς να το χρησιμοποιήσει αυτό το kit έτσι ώστε να προσαρμόσει τις ιδιαιτερότητες της κάθε χώρας αυτή την ενημερωτική εκστρατεία. Γιατί βέβαια ακόμα και αν έχουμε εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λαμβάνουν εθνικό χαρακτήρα οι εν λόγω εκλογές. Ε, και επειδή και εγώ εκλέγομαι τοπικά, αν θέλετε γνωρίζω ε, πόσο τοπικό ή εθνικό χαρακτήρα έχουν οι ευρωπαϊκές εκλογές, ακόμα και αν είναι ευρωπαϊκές. Επίσης, ε, αγγλικά, γαλλικά, πορτοκαλικά και σε κάποιες ε, άλλες χώρες, ε, νομίζω και ελπίζω και στα λιθουανικά, στη γλώσσα της Προέδρου, υπάρχει το μανιφέστο μας. Σε αυτό το μανιφέστο μπορείτε να βρείτε τις προτεραιότητές μας, οι οποίες διαθρώνονται σε, τρεις, σε συγγνώμη, πέντε ενότητες ή πέντε στόχους. Καλούμε λοιπόν για τη δημιουργία μιας συμμετοχής των γυναικών, αυξημένη συμμετοχή των γυναικών στην λήψη των πολιτικών αποφάσεων και σας έδωσα κάποια παραδείγματα προηγουμένως ως προς το τι ακριβώς εννοούμε. Επίσης απευθύνουμε μία έκκληση προκειμένου η Ευρωπαϊκή Ένωση να εγγυάται την οικονομική ανεξαρτησία όλων των γυναικών, που σημαίνει αυτό να μην υπάρχει δηλαδή ε, υψηλότερος αριθμός των γυναικών και ε, ε, γυναικείος αν θέλετε χαρακτήρας της ένδυας, αλλά και περισσότερα κοινωνικά δικαιώματα για τις γυναίκες. Επίσης, στην έκκλησή μας ζητούμε να μην υπάρχει άσκηση βίας σε βάρος των γυναικών και κοριτσιών. Πρόεδρε, αναφερθήκατε εσείς μόλις τώρα και στη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, η οποία έπαιξε το κέριο ρόλο και είναι σημαντικό κατά συνέπεια να υπογραφεί και να ακυρωθεί. Και στο πλαίσιο της επόμενης θητείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα πρέπει να υπάρξει μια οδηγία που υιοθετηθεί σε ό,τι αφορά την καταπολέμηση της βίας εις βάρος των γυναικών. Επίσης θέλουμε να έχουμε μια ε, Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία θα ε, παρέχει ασφάλεια, ειρήνη και δυνατότητες ανάπτυξης για όλες τις ε, γυναίκες. Και επίσης θέλουμε να υπάρξει κατάλληλη προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτά σε ό,τι αφορά το μανιφέστο. Αλλά τι ακριβώς ζητάμε. Βρισκόμαστε σε μια χρονική συγκυρία όπου τα δικαιώματα των γυναικών βρίσκονται το με πολλέ απειλέ, με πολλέ απειλέ επίση ενάντια στη δημοκρατία. Και είμαστε πεπισμένε ότι από κοινού μπορούμε να εμπνεύσουμε τι γυναίκε, ειδικότερα τι νέε γυναίκε, προκειμένου να έχουμε μια κοινή πρόταση ε, μια κοινή πρόταση σε ό,τι αφορά ένα κοινό μέλλον. Ένα μέλλον το οποίο θα περιλαμβάνει ακριβώς μια συμμετοχή χωρίς αποκλεισμούς αλλά και διαφοροποιημένη φιλόμορφη Ευρώπη όπου δεν υπάρχει αποκλεισμός καμίας γυναίκας και κανένας κοριτσιού. Και επίσης θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι όλες οι γυναίκες στην Ευρωπαϊκή Ένωση χαίρουν ίσων δικαιωμάτων. Και το δικό μας σλόγγαν σε αυτή την ενημερωτική εκστατεία είναι ακριβώς αυτό, η Ευρώπη για τις γυναίκες και οι γυναίκες για την Ευρώπη. Δηλαδή η Ευρώπη υποστηρίζει τις γυναίκες, αλλά θα πρέπει να το αντιληφθούν και οι γυναίκες, ότι υπάρχει αυτή η υποστήριξη και θα πρέπει να δώσουμε πραγματικά ε, νέε εναλλακτικέ μέσω αυτή τη ενημερωτική στις στι γυναίκε. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Η κυρία Λέσσα Τσεντιώνη που είναι πρόεδρος της Συμμαχίας Ευρωπαίων Γυναικών. Ευχαριστώ και ευχαριστώ που μας προσκαλέσατε για να σας παρουσιάσουμε το μανιφέστο μας. Θα ήθελα, επιτρέψτε μου, να πω δύο λόγια για την Ευρωπαϊκή Συμμαχία Γυναικών, γιατί η οργάνωσή μας δημιουργήθηκε το 2017, έχει δηλαδή μόνο δύο χρόνια ζωής, είναι μια νέα οργάνωση σε ηλικία με τη συμμετοχή όμως ε, μια ομάδας γυναικών με μεγάλο ενθουσιασμό προκειμένου ολόκληρη η κοινωνία να προχωρήσει προς ένα μέλλον με λιγότερους αποκλισμούς. Αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε την οργάνωση αυτή γιατί Αντιλαμβανόμαστε την διαδικασία που έχει αρχίσει σε πολλές χώρες ε, αποσύνθεσης ε, λίγο πολύ ε, της ευρωπαϊκής ιδέας εξαιτίας των ακραίων εθνικισμών. Εμείς λοιπόν διαπιστώνοντας ότι αυξάνεται το χάσμα το κοινωνικό σε πολλές χώρες. Ξέρουμε συγχρόνως ότι δύο είναι τα στοιχεία τα οποία υπονομεύουν τα κοινωνικά δικαιώματα και τα δικαιώματα των γυναικών και γι' αυτό και αποφασίσαμε και εμείς να αναλάβουμε δράση. Με την Ευρωπαϊκή Συμμαχία Γυναικών, λοιπόν, ασχολούμαστε με διάφορα προγράμματα. Σε ένα θέλω να επικεντρωθώ όμως κυρίως που για μας είναι το πιο σημαντικό και ε, σας καλώ να έρθετε στο επόμενο συμβούλιο μας που θα είναι εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 6 Μαρτίου είναι μια συζήτηση που γίνεται πριν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Θα έρθουν επίτροποι, ευρωβουλευτές, εκπρόσωποι από τις διάφορες χώρες μέλη, προκειμένου να συζητήσουμε την ατζέντα, του στόχους του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Υπό την οπτική γωνία βέβαια της ισότητας μεταξύ των δύο φύλων. Το έγγραφο το οποίο θα κυκλοφορήσουμε με τα συμπεράσματά μας εγκρίνεται από όσους είναι παρόντες και μετά υποβάλλεται στον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο Γιούνκερ, στον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τους και στον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ταγιάννη. Μέχρι τώρα είχαμε θετικά αποτελέσματα στη διαδικασία αυτή με μεγάλη συμμετοχή και μεγάλο ενθουσιασμό Και αυτό ακριβώς είναι και το πρώτο βήμα για μας, προκειμένου να επηρεάσουμε τη διακυβέρνηση όσον αφορά την ισότητα μεταξύ των δύο φύλων. Θέλω όμως εδώ να αναφερθώ και σε ένα άλλο Ευρωπαϊκό Μανιφέστο. Ξεκινώντας από τη βασική αρχή της οργάνωσής μας, και που είναι η καταπολέμηση των κοινωνικών αδικιών. Δεν ξέρω αν εδώ βλέπετε τη σωστή διαφάνεια ή όχι. Πιστεύουμε ότι η ισότητα μεταξύ των δύο φύλων είναι ένα βασικό στοιχείο. Δυστυχώς δεν υπάρχει ισότητα και ακριβώς αυτό είναι που πρέπει να καταπολεμήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η οικονομική κρίση του 2008 άλλαξε προς το χειρότερο την καθημερινότητα πολλών εκατομμυρίων Ευρωπαίων πολιτών. Επεριόρισε την οικονομική ανάπτυξη, την παραγωγικότητα και ενίσχυσε τους αποκλισμούς. Αυτό όμως πρέπει να αλλάξει. Να ανακτηθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών. Πρέπει να αλλάξουμε εντελώς το πρότυπο το οικονομικό και την δομή της κοινωνίας και να προτείνουμε λύσεις οι οποίες πραγματικά ανταποκρίνονται στις διεκδικήσεις του κόσμου. Γι' αυτό λοιπόν για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό το τι θα γίνει στις ευρωπαϊκές εκλογές. Εκεί πρέπει να δώσουμε την προτεραιότητα στον ηγετικό ρόλο των γυναικών και να βάλουμε τις γυναίκες στην πρώτη γραμμή που θα νομοθετήσουν. Για να το πετύχουμε αυτό λοιπόν, προτείνουμε να πάνε όσο γίνεται περισσότερες γυναίκες να ψηφίσουν στις ευρωεκλογέ. Γιατί όπως είπατε και συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Η συμμετοχή των γυναικών είναι ζωτική σημασίας για την παγίωση της δημοκρατίας και για να μεταφέρουν το μήνυμα για το ευρωπαϊκό μοντέλο που θέλουν οι γυναίκες. Εμείς προτείνουμε σε όλα τα ευρωπαϊκά κόμματα να σεβαστούν την ισορροπία μεταξύ ανδρών και γυναικών στα ψηφοδέλτια τους και να δημιουργηθεί επίσης και ένα σώμα επιτρόπων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή που επίσης να έχει ισορροπία μεταξύ ανδρών και γυναικών και γι' αυτό προτείνουμε σε όλες τις χώρες μέλη και στην κάθε μία χωριστά να προτείνουν έναν άντρα και μία γυναίκα για την κάθε θέση επιτρόπου. Οπότε όταν έρθει η στιγμή να διαμορφωθεί το σώμα των επιτρόπων να υπάρχει επιλογή να είναι εξίσου τόσο άντρες όσο και γυναίκες. Κάτι άλλο σημαντικό να αναφέρουμε εδώ είναι ότι ποτέ δεν είχαμε γυναίκα πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ή της Κεντρικής Τράπεζας ή άλλων ευρωπαϊκών θεσμών. Μόνο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που δύο φορές έχει εκλέξει γυναίκα επικεφαλής. Αυτό λοιπόν πρέπει να σταματήσει. Στην επόμενη θητεία λοιπόν εμείς θέλουμε να δούμε γυναίκες επικεφαλής των ευρωπαϊκών οργάνων. και θέλουμε μια εκπροσώπηση που να αντιστοιχεί στην πραγματικότητα. Μια άλλη πρότασή μας είναι να δημιουργηθεί ένα Συμβούλιο Υπουργών για τα δικαιώματα της γυναίκας. Τα θέματα ισότητα σήμερα συζητούνται στο Συμβούλιο ΕΣΚΟ. Όμως αυτά τα θέματα δεν συζητιούνται τόσο συχνά εκεί συχνά παραβλέπονται. Γι' αυτό επίσης θέλουμε αυτό το Συμβούλιο Γυναικών για να αποτελέσει ένα πρώτο βήμα, να δείξουμε δηλαδή προς ποια κατεύθυνση θέλουμε να πάμε. Θέλουμε οι Υπουργοί να συζητάνε για τα δικαιώματα της γυναίκας. Τώρα πηγαίνοντας προς την επόμενη θητεία, εμείς ξέρουμε ότι Φυσικά και χρειάζεται ίση εκπροσώπηση ανδρών και γυναικών, αλλά δεν φτάνει για να ενισχυθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπενθυμίζω εδώ αυτό που είπα πριν, ότι πρέπει να καταπολεμήσουμε τις κοινωνικές αδικίες. Οι επόμενοι θα πρέπει να πάρουν συγκεκριμένα μέτρα για να υπάρξουν αρκετά χρήματα στον προπολογισμό για την ισότητα ανδρών και γυναικών οι γυναίκες πρέπει να έχουν την εξουσία και τα χρήματα για να προχωρήσουν τους στόχους τους. Να υπάρχει λοιπόν ένας προπολογισμό για την ισότητα των δύο φύλων στο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο και σε όλα τα προγράμματα που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα άλλο σημαντικό θέμα για μας είναι να διασφαλίσουμε αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας σε όλες τις χώρες μέλη. Αυτό σημαίνει να υιοθετηθούν μέτρα τα οποία θα βοηθήσουν να εφαρμόζεται η αρχή ίδιος μισθός για ίδια δουλειά. Είναι και αυτό θεμελιώδης δικαίωμα. Και να διασφαλίσουμε επίσης την παιδική μέρημνα, ε, κοινωνικές υπηρεσίες για όλους, ώστε να καταπολεμηθεί ο κοινωνικός αποκλεισμός και η φτώχεια που πλήττει τις γυναίκες. Σήμερα η Οικονομική Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ψήφισε για να ορίσει δύο νέα μέλη. Ο ένας είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και ο άλλος είναι της ε, Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών. Και οι δύο άντρες. Για άλλη μια φορά λοιπόν βλέπουμε ότι οι γυναίκες δεν εκπροσωπούνται όπως θα έπρεπε σε θέσεις εξουσίας και σε διοικητικά συμβούλια. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύουμε ότι η παρουσία των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια χρειάζεται, γιατί μόνο τότε υπάρχει ισότητα και όχι μόνο αυτό. Είναι σημαντικό να υπάρχει και διαφάνεια πώς λειτουργούν τα διοικητικά συμβούλια στην ευρωπαϊκή αγορά, έτσι ώστε και οι επενδυτές να μπορούν να έχουν εμπιστοσύνη στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Ένα άλλο θέμα που θέλω να υπογραμμίσω είναι πόσο μεγάλη σημασία έχει η ψηφιακή επανάσταση. Πρέπει λοιπόν να επενδύσουμε στο ανθρώπινο δυναμικό για να πετύχει αυτή η ψηφιακή επανάσταση. Σίγουρα υπάρχει ψηφιακό χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών και μόνο αν επενδύσουμε στην διαβίου κατάρτιση και στην εκπαίδευση μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι οι γυναίκες έχουν τις ικανότητες και μπορούν να συμμετέχουν σε υψηλά επίπεδα και να μην μείνουν πίσω στην αγορά εργασίας. Τέλος, αλλά όχι και λιγότερο σημαντικό, όσον αφορά τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών. Εμείς ζητούμε στρατηγική για τη μετανάστευση για την επόμενη θητεία μια στρατηγική όπου η διάσταση του φύλου θα λαμβάνεται υπόψη. Και αυτό για να προστατεύονται τα δικαιώματα των ανηλίκων και τα δικαιώματα των γυναικών που παίζουν ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στην ε, ολοκλήρωση των κοινωνιών μας. Το μανιφέστο θα είναι έτοιμο αύριο για να μπορέσει κανείς να το υπογράψει σε όλες τις χώρες μέλη. Θα αρχίσουμε από την Ιταλία, όπου θα αποτελέσει και αντικείμενο πολιτικής εκστρατείας, που θα εγκρίνουν διάφορες γυναίκες από διάφορα πολιτικά κόμματα. Ελπίζουμε πραγματικά ότι επιτέλους οι γυναίκες θα βρεθούν στην πρώτη γραμμή αυτή τη φορά στις επερχόμενες ευρωεκλογές. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Τζεντιλόνη. Δεν θέλει κανείς το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, θέλω να κάνω κάποια σχόλια και παρατηρήσεις για κάποια σημαντικά ζητήματα που θίξατε. Οι γυναίκες είναι ίσες Είπατε πόσο δεν εκπροσωπούνται οι γυναίκες σε πολλού τομεί και κλάδου. και αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Εάν σκεφτούμε την καθημερινότητα, Τι γυναίκες να προσπαθούν να πληρώσουν λογαριασμού, να κρατάνε τον οικοκυριό, να έχουν μόνο του παιδιά, να κάνουν τρει-τέσσερι ε, διαφορετικέ δουλειέ γιατί έχουν τις συμβάσει με τις μηδενικέ ώρες και επισφαλείς θέσει. Και βλέπουμε υπέροχε γυναίκες να κάνουν θαυμάσια δουλειά και να μην πληρώνονται αρκετά. Αυτό δείχνει ότι σε όλους τους τομείς της ζωής το οικονομικό επιχείρημα ο οικονομικό ισχυρισμό ότι οι γυναίκες είναι ίσες δεν έχει φέρει αποτέλεσμα. Νομίζω είναι σαφές ότι όταν κάνουμε τα πράγματα όπως πρέπει όλοι βγαίνουν κερδισμένοι. Οι άντρε όμως ακόμα δεν πείθονται από αυτό το επιχείρημα. Δεν θα έπρεπε να είναι επιχείρημα, είναι αυταπόδεικτη αλήθεια. Πρέπει κάπως αυτό το μήνυμα να το περάσουμε, να το εκφράσουμε ακόμη πιο ηχηρά από τα σχολεία να ξεκινήσουμε. Εκεί να γίνουν οι πρώτες αλλαγές. Όταν οι γυναίκες αντιμετωπίζονται με ίσο τρόπο όλοι είναι κερδισμένοι. Αυτό πρέπει να ε, είναι ο στόχος. Να κάνουμε δουλειά για να περάσει το μήνυμα. Και να πω και κάτι για αυτό το κοινοβούλιο εδώ μέσα. Ε, ο τωρινός πρόεδρος είναι άντρας. Και το ΕΛΚ πρότεινε τη Μαρέιτ Μαγκίνες Ιρλανδή Ευρωβουλευτή. Κατά την άποψή μου, η καλύτερη ολομέλεια είναι η ολομέλεια που διευθύνει η Μαρέιτ Μαγκίνες. Εάν το σκεφτείτε από την προοπτική του Προέδρου, έχουμε μία ολομέλεια που πάει ομαλότατα, με πολλή πειθαρχία, Όλοι έχουν το χρόνο τους να μιλήσουν, έχουν και την ευκαιρία να τραβήξουν μέχρι και βίντεο. Εγώ πραγματικά πολύ λυπήθηκα που δεν μπόρεσε η Μαρέιντ να γίνει πρόεδρος του Κοινοβουλίου. Τελικά η ίδια της ομάδα την υπονόμευσε, δεν την υποστήριξε αρκετά και αυτό σημαίνει ότι οι γυναίκες δεν υποστηρίζουν τις γυναίκες οι ίδιες πολλές φορές. Στην πολιτική τα πράγματα γίνονται πολύ περισσότερο ε, εγωιστικά. Θα έπρεπε όμως να σκεφτούμε το εξή. Εάν έχουμε θέση εξουσίας, καλό θα ήταν να μην βάζουμε τρικλοποδιά σε όσου έπονται. Πρέπει να υποστηρίξουμε τις γυναίκες στους εργατικούς του labor. Έχουμε υποψήφιε γυναίκες στις περισσότερους καταλόγους υποψηφίων. Όχι για όλες τι περιπτώσει, αλλά έχει γίνει μεγάλη διαφορά γιατί αποφασίσαμε να υπάρχει ίση εκπροσώπηση των φίλων ε, στην κοινοβουλευτική μας ομάδα και γενικώ στην κοινοβουλευτική αντιπροσωπευτική δημοκρατία. Έκανε λοιπόν τεράστια διαφορά αυτό. Στου άντρε του κόμματο δεν αρέσει. Είναι σαφέ. Αλλά κερδίσαμε, ε, το πετύχαμε. Η κυρία Χάμον ήταν υπεύθυνη για αυτή την πολιτική στου ε, εργατικού. Και εγώ, ό,τι και να γίνει, θα την υπερασπίζομαι. Και αναγνωρίζω ότι οι άντρε στι ομάδε μας δεν θέλουν απαραίτητο να μας παραχωρήσουν και τη θέση τους. Είναι λοιπόν ε, μάχη πολύ μεγάλη που πρέπει ακόμα να δώσουμε. Εάν όμως μπορούμε να κερδίσουμε στο θεωρητικό επίπεδο τον αγώνα, για τα οικονομικά θέματα δηλαδή, έστω στην οικονομία που είναι κάτι το ούτω ή άλλω ηθικό, δεντολογικό, θα έπρεπε να κερδίζουμε και δεν τα καταφέρνουμε ακόμα. Γιατί η Ένωση πάντοτε κάθεται και κοιτάζει τι γίνεται στην αγορά. Αυτό τελικά είναι ο μπούσουλα. Θα πρέπει λοιπόν να τα πάμε πολύ καλύτερα για να κερδίσουμε σε θεωρητικό επίπεδο. Την αλήθεια και την πραγματικότητα την έχουμε μπροστά μας. Πώς μπορούμε να την παραγνωρίσουμε. Thank you very much. Ευχαριστούμε κυρία Γόρντ. Θέλετε το λόγο κυρία Λεφεμπρίο, κυρία Τζεντιλόνη. θέσατε τον δάκτυλο επί τον τύπο των ύλων. Είναι ακριβώς το πρώτο στοιχείο. Έτσι αποφεύγουν τη συνεργασία και αυτό είναι και το μεγαλύτερο ανυπέρβλητο εμπόδιο που ορθώνεται μπροστά μας. Οι λόγοι είναι λόγοι νοοτροπίας. Εμείς ως γυναίκες πρέπει ακόμα να κάνουμε πολλή δουλειά για να ξεπεράσουμε αυτούς τους περιορισμούς. Όμως, εκτός που πρέπει να συνεργαστούμε για να δικτυωθούμε μεταξύ μας και να περάσει ένα μήνυμα αλληλεγγύης και φεμινισμού και αμοιβαίας συνεργασίας, πρέπει να πω ότι χρειάζεται χρόνος. Χρειάζεται χρόνος και από την προσωπική μου εμπειρία, από τη δουλειά μου σε αυτή την οργάνωση, πρέπει να πω το εξής. Όταν οι γυναίκες φτάνουν σε θέσεις κορυφαίες, δεν υποστηρίζουν αναγκαστικά άλλες γυναίκες ή δεν υποστηρίζουν τον σκοπό μας. Είναι ευκολότερο για κάποιον να πάει στην παράταξη των ε, γυναικών για να προχωρήσει ο αγώνας μας, αλλά δεν γίνεται πάντοτε έτσι. Θα συμφωνήσω λοιπόν με την κυρία Γόρντ, ε, πρέπει να κερδίσουμε ό,τι και να γίνει και γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε σε στενή συνεννόηση και συνεργασία. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Λαφαμπρία. Ευχαριστώ. Αναφέρατε πολλά ζητήματα στην παρέμβασή σας. Πρώτα απ' όλα, γιατί να ψηφίσει ο κόσμος φεμινιστές στις επόμενες εκλογές. Γιατί να το θέλουμε αυτό. Όταν λέμε φεμινιστές, δεν εννοούμε γυναίκες. Φεμινιστές άντρες θέλουμε. Συμφωνούμε νομίζω. Γι' αυτό υποστηρίζουμε ψήφο υπέρ των γυναικών και υπέρ των φεμινιστών ε, υποψηφίων. Παντού στην Ευρώπη θέλουμε να στηρίξουμε φεμινιστές υποψηφίου, την άντρε ή την γυναίκες. Αυτό είναι δεδομένο. Είπατε πώς μπορεί να χτιστεί η ισότητα, η ισοτιμία σε όλες τις κοινωνικές εκφράσεις, τα σχολεία, ε, την οικονομία. Να σας αναφέρω ένα παράδειγμα που το γνωρίζω καλύτερα. Ο νόμος περί στη Γαλλία πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε την εκλογή περισσότερων γυναικών βάσει ενός νόμου για την ισότητα. Διότι σε όλες τις εκλογές πλέον υπάρχει ισότης. Δεν είναι το μόνο, είναι όμως ένας τρόπος να επηρεαστούν οι νοοτροπίες και να προβάλλουμε τα κατάλληλα πρότυπα Ανθρώπου πρότυπα γιατί αυτό που χρειαζόμαστε για τι γυναίκες και τα νερά, τα νερά κορίτσια και τι νεαρές γυναίκες είναι να τους δείξουμε συγκεκριμένου συγκεκριμένους ανθρώπους ως πρότυπα να τους δείξουμε ότι και εσύ έχεις τις γνώσεις και τις δεξιότητες και μπορείς να τα καταφέρεις γιατί αυτά δεν προβάλλονται στις οθόνες του στα κοινωνικά δίκτυα Όπω το είπατε για την πρόεδρο του Κοινοβουλίου, τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου. Εάν δει κανεί, ε, αν δει κάποια κοπέλα, μια άλλη γυναίκα ότι τα καταφέρνει, ε, ενθαρρύνεται. Είναι ένας τρόπος να ταυτιστεί. Αυτό λοιπόν θα μπορούσε να επιτρέψει να, έχουμε, να ξεκινήσει μάλλον να έχουμε ισότητα ή εκπροσώπηση στους εκλογικούς καταλόγους, ε, στη, στα ψηφοδέλτια μάλλον, των κομμάτων μας ήδη. σε εκπροσώπηση ανδρών και γυναικών. Και είναι καλό και για τους δύο, και για τους άντρες και για τις γυναίκες. Διότι οι άντρες σε ένα φεμινιστικό περιβάλλον δεν χρειάζεται να ε, φορτωθούν το βάρος της τοξικής παρουσίας υπερβολικά πολλών ανδρών. Οι άντρες μόνοι τους αφήνονται και εκφράζονται όπως να είναι. Ξεκινά από το σχολείο αυτό. Οι γυναίκες καλό να είναι παρούσες σε όλες τις φάσεις της ζωής τους να ξεκινήσουμε να εργαζόμαστε από το σχολείο και μετά και στο κοινοβούλιο, τα πολιτικά κόμματα όπως είπατε. Και αυτά είναι καλές αφορμές. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Λαφευρία. Και τώρα να ευχαριστήσω και τις δυο σας και τις δύο οργανώσεις, το λόμπι των γυναικών και το λόμπι Αλιανς, για τις πρωτοβουλίες σας, για όλα αυτά που κάνετε. Πραγματικά μας βοηθάτε ως πολιτικούς να πετύχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Χρειαζόμαστε περισσότερε γυναίκε στο Ευρωκοινοβούλιο και στι Εθνικέ Βουλέ, στι αρχέ Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Πολύ σα ευχαριστώ. Και νομίζω ότι με τη συνεργασία μα θα πετύχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Ευχαριστώ πολύ. Θα κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα έως τις 5, ε, οπότε και θα συνεχίσουμε. Και στι 5 θα ξεκινήσει η ψηφοφορία. Συνάδελφοι, ας ξεκινήσουμε την ψηφοφορία μας. Έχετε όλοι τις ε, κάρτες σας να ξεκινήσουμε. Περνάμε λοιπόν στο σημείο 6 της ημερήσιας διάταξης. Θέσπιση κανόνων για τη στήριξη των στρατηγικών σχεδίων που πρέπει να καταρτίζονται από τα κράτη-μέλη στο πλαίσιο τη κοινή γεωργική πολιτική και να χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτική Ανάπτυξη. Η Μαριάννα Πετήρη είναι η συντάκτρια του τη γνωμοδότηση και θα ξεκινήσουμε την ψηφοφορία λοιπόν τώρα. Τροπολογία 31 υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα πρέπει να ελέγξουμε την 39 ηλεκτρονικά. άρχιτη ψηφοφορία. Υπάρχει μία ψήφος παραπανέσια από την πλευρά του ΕΛΚ. Now it's okay, yeah? The vote is closed. It's adopted. Εγκρίνεται. Τροπολογία 40 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 41 υπέρ. Θέλετε να ελέγξουμε τροπολογία 40 πρώτα. Καλώς ελέγχουμε ηλεκτρονικά άρχη ψηφοφορία. Πέραση της ψηφοφορίας εγκρίνεται. Με την ίδια πλειοψηφία, όπως και 39. Περνάμε στην τροπολογία 41 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 1 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 42 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 43 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Όχι, δεν χρειάζεται να ελέγξουμε γιατί ήταν ε, σαφές το αποτέλεσμα από την αντίθεση. 44 λοιπόν σε δύο μέρη. Πρώτο τμήμα υπέρ. Α, όχι καταπίπτει το πρώτο ε, τμήμα της γιατί έχει εγκριθεί η συμβαστική τροπολογία 1 οπότε περνάμε στο δεύτερο τμήμα 44 επερ κατά αποχές εγκρίνεται. Ας ελέγξουμε όμως. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Πέρας. Εγκρίνεται. 46 τώρα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 2 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 49 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 51 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 52 υπέρ, όχι, ας ελέγξουμε ηλεκτρονικά την τροπολογία 51. Ξεκινάμε λοιπόν, άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Ή μάλλον έχει καταπίψει. Οπότε 52 υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα πρέπει να ελέγξουμε την τροπολογία 52. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. απορρίπτεται. 53 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 3 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 56 τώρα. Πρώτο τμήμα. Α, όχι, έχει καταπίπτει το πρώτο τμήμα της 56, ε, αλλά και το δεύτερο τμήμα της 56 ε, καταπίπτει. Οπότε περνάμε στη συμβαστική τροπολογία 4 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 57 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 61 υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα ελέγξουμε την τροπολογία 61. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 62 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 63 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 60 5 υπέρ κατά αποχές θα ελέγξουμε την 65 ηλεκτρονικά άρχεται ψηφοφορία πέρας εγκρίνεται συμβαστική τροπολογία 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 68 υπέρ κατά αποχές θα ελέγξουμε την 68 ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 69 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται με την ίδια πλειοψηφία. Συμβασική τροπολογία 6 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβασική τροπολογία 7 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 73 υπέρ α όχι 71 μαζί με την 116 από κοινού υπέρ κατά αποχές θα πρέπει να ελέγξουμε αυτές τις δύο τροπολογίες 71 και 116 άρχεται η ψηφοφορία πέρας εγκρίνονται. 72 υπέρ κατά άποχες με την ίδια πλειοψηφία εγκρίνεται και 72 περνάμε στην 73 υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται 74 υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται 75 υπέρ κατά αποχές ας ελέγξουμε την 75 ηλεκτρονικά άρχεται ψηφοφορία πέρας απορρίπτεται τροπολογία 76 σε δύο τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές Εγκρίνεται. Τώρα, 77, 100 και 85, αυτές οι τροπολογίες από κοινού υπέρ, κατά, αποχές, θα πρέπει να τις ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτονται. 79 υπέρ κατά αποχές Ας ελέγξουμε την 79 ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Ε, Amendment 81. 81. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 82 υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα πρέπει να ελέγξουμε την τροπολογία 82 ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα τη ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 83 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 84 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε την 84 ηλεκτρονικά άρχη της ψηφοφορία πέρας εγκρίνεται Συμβαστική τροπολογία 8. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 86 υπέρ, κατά, αποχές. Θα ελέγξουμε τροπολογία 86 ηλεκτρονικά. Άρχεται ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 9 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 94 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 95 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 96 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Να ελέγξουμε όμως ε, την 96, ε, ηλεκτρονικά έρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Η συμβαστική τροπολογία 11 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 98 υπέρ. Κατά θα πρέπει να ψηφίσουμε από τις 98 υπέρ, κατά, αποχές. Θα ελέγξουμε λοιπόν την 98, άρχη ψηφοφορία. The vote is closed. Απορρίπτεται λοιπόν. Περνάμε στην τροπολογία 101. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ε, ζητώ συγγνώμη, ε, συνάδελφοι, θα πρέπει να ψηφίσουμε και επί της 97 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Να ελέγξουμε όμως την 97 ηλεκτρονικά, άρχεται ψηφοφορία. Πέρας, εγκρίνεται. Περνάμε στη συμβαστική τροπολογία 12 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 106 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 107 υπέρ, Now we are now. Συνάδελφοι, πρέπει να ψηφίσουμε τις 105, τροπολογία 105. Είναι πολύ περίπλοκα τα πράγματα. Σα ζητώ συγγνώμη. Συγγνώμη, είναι αυτό ο κατάλογο ψηφοφορία λίγο περίπλοκο. Γιατί πρέπει να ψηφίσουμε ω προσθήκη στην συμβαστική τροπολογία 12 την 105. Υπέρ λοιπόν τη 105. Κατά αποχέ θα ελέγξουμε την 105 ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Απορρίπτεται. Τώρα περνάμε στην 107 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Να την ελέγξουμε όμως ηλεκτρονικά. Την 107, άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 14, υπέρ, κατά, αποχές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 113 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 115 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 117 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 118 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 13 υπέρ, κατά, αποχές, εκρίνεται. Τροπολογία 21 υπέρ, κατά, αποχές, θα πρέπει να ελέγξουμε την τροπολογία 21 ηλεκτρονικά, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Τροπολογία 24 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 25 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 2 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 27 υπέρ, κατά, εποχές, εγκρίνεται. 30 υπέρ, κατά, εποχές, εγκρίνεται. Να κάνουμε έλεγχο για τα 30. Εγκρίνεται. 29 υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 31 πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Δεν, χρειάστηκε να, δεν χρειάζεται να ψηφίσουμε τα 31. Συγγνώμη, συναδελφοί. Καταπίπτει. Κατέπεσε δηλαδή. Πάμε στην 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 32. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 33. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι εγκρίνεται, αλλά καλύτερα να ελέγξουμε. Ας ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Η 34 καταπίπτει. Πάμε στα 36 υπέρ. Κατά. Αποχές. Συνάδελφοι, σηκώνετε παρακαλώ τα χέρια σας. 36 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 35 35 καταπίπτει. 5 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 6 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 37 υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. 38 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Και τώρα το σχέδιο της νομοδότησης ως τροποποιήθηκε, ονομαστική κλίση, άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας. Συγχαρητήρια στην εισηγήτρια, κυρία Πετήρ και σε όλους τους κοιόδους εισηγητές. Πολύ σας ευχαριστούμε. Κυρία Πετήρ Μαριάννα, θέλετε το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συνάδελφοι, να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία για να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους και ευρωβουλευτές που επέτρεψαν να έχουμε αυτήν την ε, πολύ καλά εξισορροπημένη γνωμοδότηση για τα στρατηγικά προγράμματα των κρατών μελών σε σχέση με την ΚΑΠ. Υπήρχε μεγάλη σύγχυση για την σχετική αναθεώρηση. Ευχαριστώ ιδιαίτερα τους συναδέλφους από την ομάδα του ΕΛΚ που πραγματικά υποστήριξαν τις περιοχές της Υπέθρου και τη Γεωργία για να έχουμε υψηλής ποιότητας ΚΑΠ. Αναζητούμε τρόπους να δώσουμε περισσότερες δυνατότητες στις γυναίκες που εργάζονται στην Υπέθρου. Δεν θέλουμε να τις φορτώσουμε με επιπλέον βάρος ε, διοικητικό. Πρέπει να υπάρχει σωστή ισορροπία της δουλειάς ανδρών και γυναικών στα αγροτικά. Ε, γι' αυτό απλώς θέλουμε να είναι ομαλότερη η εφαρμογή της ΚΑΠ στα κράτη-μέλη. Ως εισηγήτρια και μέλος της Επιτροπής Άγκρη θα φροντίσω να λάβω τα απαραίτητα μέτρα, την απαραίτητη μέρημνα, για να φτάσει αυτό στην αρμόδια επιτροπή. Σκοπός είναι να δώσουμε περισσότερες δυνατότητες, να βοηθήσουμε τις γυναίκες της επέτρου να χειραφετηθούν. Thank you. Thank you. And now... Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε στο επόμενο σημείο στην ημερήσια διαταξή. Σημείο 7. Ο ρόλο των γυναικών στην πρόληψη τη ριζοσπαστικοποίηση. Η κυρία Χιμένες Μπεσερίλ Μπάριο. Να ψηφίσουμε τώρα ηλεκτρονικός. Η Γκούε και η Πράσινοι ζήτησαν κάτι όμως. Ναι, ναι, κυρία Μπιόρκ, μάλλον. Συνάδελφοι, είναι πραγματικά μια συνήθιστη έκκληση να ζητηθεί η αναβολή της ψηφοφορίας για την Επιτροπή μας και πιστεύουμε ότι θα μπορούσε να βελτιωθεί πάρα πολύ η έκθεση. Η κοινωνία των πολιτών εκτός του Κοινοβουλίου μας έχει ειδοποιήσει ότι το ψήφισμα αυτό δεν είναι καθόλου σωστά εξισορροπημένο και θέλουν να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να ε, προλάβουμε τη ριζοσπαστικοποίηση, που δεν γίνεται με την τροπή που έχει πάρει το ψήφισμα. Πολλά πράγματα. Ο στιγματισμό ομάδων γυναικών, ιδίω των ε, μουσουλμάνων. Δεν ασχολείται ε, με τις ακραίες μορφές ριζοσπαστικοποίησης. Πρέπει να μιλήσουμε και για το συγκεκριμένο φαινόμενο το μανιφέστο 36 που ήταν ε, ιδιαίτερα στοχευμένο πρέπει να προστατεύσουμε όλες τις κοινότητες που του ε, ψηφίσουμε για το θέμα αυτό. Θα ζητούσαμε λοιπόν την αναβολή της ψηφοφορίας έως τις 2 Απριλίου. you, Ms. Ευχαριστούμε κυρία Μπιόρκ. Η κυρία Χιμένες Μπεθερίλ. Ευχαριστώ. Πρέπει να σας πω ότι με εκπλήσει το αίτημα αυτό που μου φαίνεται ότι δεν στέκει τη στιγμή που έχουμε λάβει 103 τροπολογίες για τις οποίες ευχαριστώ. Οι περισσότερες είναι μια επανάληψη και βρίσκονται εκτός του πνεύματος του ψηφίσματος αυτού. Προσπαθήσαμε όμως να κάνουμε διαπραγματεύσεις, καταλήξαμε σε πέντε συμβιβαστικές, έχουμε ανταλλάξει διάφορα email, κανείς δεν ζήτησε κάποια επιπλέον συνάντηση, οπότε δεν αντιλαμβάνομαι το αίτημα αυτό για αναβολή. Έχουμε από το Δεκέμβριο που αρχίσαμε να δουλεύουμε πάνω σε αυτό το κείμενο. Υπενθυμίζω ότι δεν πρόκειται ούτε για οδηγία ούτε για κανονισμό, πρόκειται για ένα ψήφισμα για ένα θέμα που εγώ προσωπικά ζήτησα. Είναι δικιά μου έκθεση αυτή. Ψηφίστηκε στους συντονιστές. Έπειτα το πνεύμα, το λέω, γιατί με αυτό το πνεύμα ακριβώς ζητήσαμε ε, το κείμενο αυτό, κάναμε πάρα πολλές ακροάσεις για την ριζασπαστικοποίηση των γυναικών Έχουμε συναντηθεί με μητέρες, με το διευθυντή για την τρομοκρατία, ε, με γονείς ε, ριζοσπαστικομένων νεαρών που λένε ότι χάρη στα προγράμματα οι γυναίκες μπορούν να βοηθούν τα αγόρια αυτά. Συναντηθήκαμε με γυναίκες που έχουν παιδιά που έρχονται από τη Συρία και θέλουν να ενταχθούν και πάλι τα παιδιά αυτά και οι, όχι μόνο οι γονείς και οι γιαγιάδες ακόμα αυτών των νεαρών θέλουν να βοηθήσουν στην επανένταξή τους στην κοινωνία. Εγώ προσωπικά το έχω πει σε πολλούς ανθρώπους, έχω δώσει πολλές συνεντεύξεις και με τίποτα το ψήφισμα αυτό δεν είναι ανώριμο κάθε άλλο. Ούτε στιγματίζει κανέναν. Αν δείτε τις εντρολογικές σκέψεις, τι έγινε στην Επιτροπή Διαλόγου, είδε γυναίκες από την Επιτροπή της Μεσογείου, όλοι αυτοί λένε ότι πρέπει να βοηθήσουμε τους νέους που βρίσκονται είτε στη Στέουτα και στη Μελίγια Ιταλού και βλέπουν ότι μπορεί κανείς μέσω της προπαγάνδας στο διαδίκτυο να ενταχθούν σε τρομοκρατικά δίκτυα. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύω ότι πέρα από το ότι η διαδικασία ήταν ξεκάθαρη, με διαφάνεια, με τις τροπολογίες της, τώρα το μόνο που μας μένει είναι να ψηφίσουμε. Συνεπώς, εγώ δεν συμφωνώ να αναβληθεί η ψηφοφορία. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Πεθερίλ. Δεν χρειάζεται να το συζητήσουμε περαιτέρω, θα ψηφίσουμε. Για το αίτημα Γκούε και Πρασίνων, για αναβολή. Αναβολή για το προφορικό ερώτημα και το ψήφισμα. Η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. We vote on the request to Ψηφίζουμε το αίτημα αναβολής. is too much. Υπάρχει ένας παραπάνω από ό,τι θα έπρεπε. Τώρα είμαστε εντάξει. Πέρας. Απορρίπτεται. Οπότε ψηφίζουμε κανονικά. προφορική ερώτηση, πρόληψη των, ε, της συμμετοχής των γυναικών στη ριζοσπαστικοποίηση. Τροπολογία 1. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Θέλετε έλεγχο για την πρώτη τροπολογία, να ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφορία. Τροπολογία 1. Πέρας. Απορρίπτεται. 2. Υπέρ. Κατά. Εποχές. Έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία. Συνάδελφοι, τελική ψηφοφορία για το κείμενο της προφορικής ερώτησης όπως διορθώθηκε. Ηλεκτρονική. Τελική ψηφοφορία. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια. Και τώρα επόμενο σημείο. Συνάδελφοι, τώρα θα ψηφίσουμε το ψήφισμα ρόλο των γυναικών στην πρόληψη τη ριζοσπαστικοποίηση τη κυρία Τερέζα Χιμένε Μπεσερίλ Μπάριο, να σα ενημερώσω ότι ω προ την ψηφοφορία για το ψήφισμα ενημερωθήκαμε σήμερα το απόγευμα ότι λόγω διοικητικού προβλήματος οι τροπολογίες που αρχικά είχαν υποβληθεί από τους συντηρητικούς και μεταρρυθμιστές δεν συμπεριελήφθησαν στο έγγραφο των τροπολογιών. Για το λόγο αυτό θα υποβληθούν προφορικώς. Σας δίνουμε το λόγο να παρουσιάσετε αυτές τις ε, προφορικές τροπολογίες. Όταν θα έρθει η στιγμή στην κατάλληλο ψηφοφορία. Αρχίζουμε να ψηφίζουμε για το ψήφισμα. Αυτό σημαίνει ότι θα διαβάζουμε μόνο το κείμενο το οποίο θα ψηφίζουμε. Μα τώρα σοβαρός είναι απαράδεκτο από άποψη διαδικασία. Και δεν είναι και δίκαιο για του άλλου συναδέλφου. Εγώ δεν τι έχω δει αυτέ τι τροπολογίε και δεν είμαι καθόλου έτοιμη να ψηφίσω από αυτόν. Δεν γνωρίζω καν καλά το κείμενο. Θέλω τουλάχιστον να έχω μπροστά μου το κείμενο τυπωμένο. Uh, Miss Κυρία Ρέντκε, είναι διοικητικό το πρόβλημα, καταλάβατε. Οι τροπολογίες αυτές υποβλήθηκαν ε, γέρος. Και τώρα θα σας τις δώσουμε και γραπτός. Από τους κλητήρες θα τις λάβετε. Ναι, κυρία Μούντι, ευχαριστώ. Κοιτάξτε, καταλαβαίνω τη δυσκολία από την άποψη τη διοργανωτική. Είναι διοικητικό, ωραία, δεν θέλουμε να κατηγορήσουμε κάποιον προσωπικά. Όμω, αντικειμενικά η δουλειά μα είναι να ψηφίσουμε πράγματα τα οποία ε, τα έχουμε αποφασίσει βάσει τεκμηριωμένη εξέταση ενό κειμένου. Δεν μπορούμε εντελώ όμω ειλικρινά και με το χέρι στην καρδιά να πούμε ότι έχουμε τώρα την δυνατότητα να, έχουμε να λάβουμε μια απόφαση τεκμηριωμένη. Δεν υπάρχει λόγο να κατηγορηθεί κανεί. Είναι πρόβλημα. Είναι αντικειμενικά πρόβλημα. Ω νομοθέτε δεν μπορούμε να παίζουμε. Δεν μπορούμε να το δεχτούμε ω ε, επί τη αρχή. Συγγνώμη και από μένα. Κοιτάξτε. Είπε η γραμματεία ότι υπήρξε τεχνικό πρόβλημα της γραμματείας πριν από λίγο η Πρόεδρος είπε ότι υπάρχει δυνατότητα όταν υπάρχει τεχνικό ζήτημα δεν είναι τροπολογίες της τελευταίας στιγμής, δεν είναι κάτι πολιτικό, ούτε μιας πολιτικής ομάδας, ούτε τίποτα. Πρόκειται για τροπολογίες οι οποίες είναι όπως πρέπει, αλλά περνώντας από το Word σε ένα άλλο σύστημα δεν πέρασαν. Και αυτό έγινε αντιληπτό εδώ και η πρόεδρος η οποία έχει τη διακριτική δυνατότητα, είπε ότι εφόσον πρόκειται για τεχνικές τροπολογίες, μπορούμε να τις ψηφίσουμε. Άλλο είναι να μην θέλει κάποιο να ψηφίσει την έκθεση αυτή, αλλά καμιά σχέση με αυτή τη τεχνική φύσεω τροπολογίε. Παρακαλώ. Κοιτάξτε, εγώ δεν θα μπω τώρα στο θέμα του κατά πόσο είναι τεχνική φύσεω ή όχι τροπολογίε, γιατί όπω είπε και η συνάδελφο, δεν πρόκειται εδώ να ψάξουμε να βρούμε ποιος φταίει. Αν υπάρχει δεν υπάρχει ευθύνα. Ε, πήρε το λόγο. Τώρα η σειρά μου. Μην με διακόπτεις. Τώρα μιλάω εγώ. Λοιπόν, εμάς ε, θέλετε να μας βάλετε να ψηφίσουμε διάφορες τροπολογίες που μόλις τώρα πήραμε στα χέρια μας. Να τις ψηφίσουμε ή ε, όχι. Είναι πρωτοφανές. Μπορεί να ήταν τεχνικό το πρόβλημα, Δώστε μας λίγο χρόνο. Κάτι. Ε, πραγματικά. Είμαστε όλοι υπεύθυνοι όταν ψηφίζουμε. Η ψήφος είναι κάτι σημαντικό. Δεν μπορεί κανείς να πηγαίνει και να ψηφίζει έτσι χωρίς να το έχει δει πριν και χωρίς να ξέρει περί τίνος πρόκειται. Δεν είναι τεχνικά αυτά τα ζητήματα. Εδώ πέρα βλέπω ότι μιλάει για το ISIS. Όχι, όχι, καθόλου. Εγώ δεν πρόκειται να ψηφίσω. Αρνούμε να το ψηφίσω εγώ αυτό. Κοιτάξτε, πρόκειται για προφορικές τροπολογίες. Είναι ένα τεχνικό το ζήτημα από την αρχή, σύμφωνη, αλλά καταλήγει να γίνεται πολιτικό, γιατί πρόκειται για τροπολογίες ε, οι οποίες δεν μας βρίσκουν σύμφωνους και δεν έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε μεταξύ μας. Συνήθως καθόμαστε, διαπραγματευόμαστε, εδώ δεν ξέρουμε. Γι' αυτό κι εγώ είμαι κατά ε, των προφορικών αυτών τροπολογιών. Καταλαβαίνω ότι καταρχήν είναι τεχνικό το ζήτημα, αλλά καταλήγει να γίνεται πολιτικό κάτω από αυτές τις συνθήκες. Ε, Πρόεδρε, οι συνάδελφοι, οι τροπολογίες αυτές είναι πάρα πολύ απλές. Είναι όλες σύντομες και ε, παραλαμβάνουν μέρη του κειμένου που είχαν διαγραφεί. Νομίζω ότι με ένα τεχνικό διάλειμμα 5 λεπτών προλαβαίνετε να τις δείτε όλες. Είναι ελάχιστες φρασούλες στο κείμενο, μέρος του κειμένου που είχε διαγραφεί. Τίποτε άλλο. Very quick. If I Επιτρέψτε μου πολύ σύντομα να πω κάτι. Όταν λέτε είναι τεχνικό, δεν είναι και το επαναλαμβάνετε αυτό, εγώ ξέρω και το λέει πρόεδρος ότι υπάρχει ένα τέχνικο. Το λέω και εγώ ότι είναι τεχνικό, αλλά επειδή το λέει η πρόεδρος και το επιβεβαιώνει και η γραμματεία ότι υπήρξε ένα τεχνικό πρόβλημα. Είχαν υποβληθεί. Αν δεν είχαν υποβληθεί, εντάξει. Αλλά εδώ δεν έγινε κάτι στραβό. Είναι καθαρά τεχνικό το ζήτημα είναι πρόβλημα που προέκυψε στην γραμματεία. Προσπαθούν να το λύσουν στη γραμματεία με τον καλύτερο τρόπο και την καταλαβαίνουν τη γραμματεία. Είναι ένα τεχνικό ζήτημα, οπότε δεν πρέπει να δώσουμε παραπάνω βάρος. Εφόσον το λέει και η Πρόεδρος, το υπόσχεται Now five minutes break. Πέντε λεπτά διάλειμμα. Κατά τη διάρκεια του διαλύματος θα διαβάσετε. Διαβάστε τις τροπολογίες και μετά θα ψηφίσουμε. Και αν δεν συμφωνείτε με τις τροπολογίες, να τις καταψηφίσετε. Καταψηφίστε τες. Θα ξεκινήσουμε μετά από 5 λεπτά. Uh, Αγαπητοί συνάδελφοι, θα συνεχίσουμε. Ψηφίζουμε λοιπόν. Αρχίζουμε να ψηφίζουμε και θα ψηφίσουμε την τροπολογία 67 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 68 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Θα ελέγξουμε καλώς. 68. Μπορείτε να ψηφίσετε. Τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. Τροπολογία 69 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 70 υπέρ, κατά, αποχές, θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίστε. Τέλος.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 κατά, αποχές, εγκρίνεται. 77 υπέρ, κατά, αποχές, θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά για την 77. Ψηφίστε παρακαλώ. Τέλος της ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε. 78 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 79 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 80 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 81 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 82 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 83 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 84 υπέρ, κατά, αποχές, θα ελέγξουμε την 84 ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ. Τέλος της ψηφοφορίας.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 θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά για την 89. Ψηφίστε παρακαλώ. Τέλος της ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε. Τροπολογία 90 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 91 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά για το δεύτερο τμήμα. Ψηφίστε παρακαλώ. Τέλος της ψηφοφορίας. Απορριφθήκε το δεύτερο τμήμα. 92 τροπολογίες σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 93 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 94 υπέρ, κατά, αποχές, θα Α, εγκρίθηκε, εγκρίθηκε. Τροπολογία 95 τώρα. Υπέρ. Ψηφίζουμε για τη διαγραφή. Υπέρ λοιπόν. Κατά. Νομίζω ότι απορρίπτεται, αλλά σε ελέγξουμε καλύτερα. 95. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε. Τώρα, ε, τροπολογίες PCR. Ποιος θα τις διαβάσει. 4. Αριθμός 4 του ECR. Από αυτές που κατατέθηκαν στο έγγραφο τροπολογιών. Κύριε Γκέρκε, ακούμε. Ίσως δεν χρειάζεται, γιατί τις ξέρετε, έτσι δεν είναι. Τις έχετε, τις έχετε γραπτά. Οπότε δεν χρειάζεται να τις διαβάσουμε. Ωραία. Ψηφίζουμε τροπολογία αριθμός 4 του ECR. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Απορρίφθηκε. Τροπολογία 96 τώρα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίφθηκε. 97 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 98 υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. 99 υπέρ, κατά, αποχές, θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά για την τροπολογία 99. Ψηφίστε παρακαλώ. Τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. Τροπολογία 100 υπέρ, κατά, αποχές, θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά για την 100. Ψηφίστε παρακαλώ. Τέλος της φοφορίας. Απορρίφθηκε. Τροπολογία 101 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 102 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 103 υπέρ. Κατά. Αποχές θα ελέγξουμε για την 103 ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ. Τέλος της φοφορίας. Απορρίφθηκε. 104 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 105 υπέρ. Κατά. Αποχές. 105 υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ. Τέλος της φοφορίας. Απορρίφθηκε. 106 τώρα υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 107 υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά για την 107. Ψηφίστε παρακαλώ.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 26 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 27 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 29 υπέρ, κατά. Α, 28, ναι, διορθώνει η πρόεδρος, συγγνώμη, 28 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 29 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 30 υπέρ, κατά, αποχές, θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά για την 30, ψηφίστε παρακαλώ. Τέλος της ψηφοφορίας και απορρίφθηκε. 31 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 32 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 1 υπέρ, κατά, αποχές, Εγκρίνεται. 36 τώρα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Και τώρα η τροπολογία αριθμός 1 του ECR υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 37 υπέρ. Κατά. Αποχές. πρέπει να ελέγξουμε για την 37. Ψηφίστε παρακαλώ ηλεκτρονικά. Τέλος της φοφορίας Απορρίφθηκε. 38 υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα ελέγξουμε. 38. Ψηφίστε παρακαλώ. Τέλος της φοφορίας Εγκρίθηκε. Τριάντα εννέα τώρα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Σαράντα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Σαράντα ένα υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά για τη 41. Ψηφίστε παρακαλώ. Τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. 42 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 43 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 45 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 46 υπέρ, κατά, αποχές, θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά για τη 46. Ψηφίστε παρακαλώ. Τέλος της ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε. 47 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τώρα, τροπολογία αριθμούς 2 του ECR υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 48 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 49 υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. 50 υπέρ, κατά, αποχές, θα ελέγξουμε. Ψηφίστε παρακαλώ ηλεκτρονικά για την 50. Τέλος της φοφορίας. Απορρίφθηκε. 51 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 52 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 53 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 54 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 55 υπέρ κατά αποχές θα ελέγξουμε για την 55 ηλεκτρονικά. Μπορείτε να ψηφίσετε. Τέλος της ψηφοφορίας και απορρίφθηκε. 56 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τώρα, τροπολογία 3 του ΙΣΙΑΡ. Υπέρ παρακαλώ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 57 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται.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 κατά, αποχές, εγκρίνεται. 13 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Α, θέλετε να ελέγξουμε. Ωραία, για τη 13. Μπορείτε να ψηφίσετε. Τέλος της ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε. Με μια ψήφο διαφορά, ναι. 14 υπέρ, κατά, αποχές, θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ.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 το τροποποιημένο ψήφισμα ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε. And, and now the vote is closed. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. Συγχαρητήρια στην εισηγήτρια κυρία Μπεσερίλ Μπάριο. Μάλιν. στην συνεδρία των συντονιστών αποφασίστηκε να μην περάσει το ψήφισμα αυτό στην Ολομέλεια. Ελπίζω να το σεβαστούν όλες οι ομάδες. Θα ήθελα όμω να επισημάνω ότι θέλω να υποβάλω ένα ψήφισμα μειονοτικό εξ ονόματος της Επιτροπής. Μπορείτε να το προσθέσετε στα πρακτικά. Ε, δείτε αν είναι εφικτό. Ούτως ή άλλως σήμερα παρεβήκαμε πολλές φορές του μεσοτρικό κανονισμού. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, καλή ψηφοφορία, αλλά περίπλοκη. Χρονοδιάγραμμα, δύο λεφτά. Πρέπει να ψηφίσουμε. Α, να προσαρμόσουμε το χρονοδιάγραμμα. Δεν βλέπω να υπάρχουν αντιρρήσεις. Εγκρίνουμε. Τελείωσε η ψηφοφορία και πάμε στο τελευταίο σημείο Yes, we have Έχουμε λοιπόν ένα ακόμα σήμερα στην ημερήσια διάταξη. Η κυρία Γνιέστα Κοσλόφσκα θα μας παρουσιάσει. Είστε έτοιμοι να πάρετε το λόγο. Σε σχέση με αυτό το επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξη, το 9, ε, η τριμερής διάλογη σχετικά με την ισορροπία μεταξύ επαγγελματική και ιδιωτική ζωής. Παρακαλώ λοιπόν, Αγνιάσκα, ω εισηγήτρια μπορείς να πάρει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε θα αξιοποιήσω την ευκαιρία να μιλήσω στα πολωνικά που είναι με τέτοιου μου γλώσσα, οπότε αν θέλετε βάλτε τα ακουστικά σας ε, για να με ακούσετε. Γιατί δεν νομίζω ότι μιλούν πολύ στην αίθουσα. E, Καταρχήν, θα ήθελα να εκφράσω την ικανοποίησή μου για το γεγονός ότι η εν λόγω πρόταση σε ό,τι αφορά την ισορροπία μεταξύ επαγγελματική και ιδιωτική ζωή έχει προταθεί από δύο Επιτρόπους και πλέον έχουμε φτάσει στην οριστική κατάληξη σε ό,τι αφορά αυτό το φάκελο. Επρόκειτο για ένα δύσκολο ζήτημα, αλλά εμείς από την πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υπήρξαμε φιλόδοξοι. Θέλαμε δηλαδή ε, να διασφαλίσουμε ότι υπάρχει υψηλή αμοιβή ε, σε ό,τι αφορά την γονική άδεια Ωστόσο είχε ε, απορρίψει το Συμβούλιο μια ε, πρόταση αυτού του είδους γιατί οι απόψει των κρατών μελών ήταν εντελώ διαφορετικέ από αυτές του Κοινοβουλίου. Άρα λοιπόν ήταν δύσκολες οι διαβουλεύσεις και δύο φορέ φτάσαμε σχεδόν στο, στη διακοπή των διαβουλεύσεων. Και κατά τη διάρκεια όλη αυτή τη διαπραγμάτευση ε, το Συμβούλιο μα προσέγγισε σε πολύ μικρό βαθμό. Ε, έδειξε δηλαδή μικρή ευελιξία και έτσι το τελικό αποτέλεσμα εδώ δεν είναι εκείνο που εμείς ευχόμασταν να έχουμε στην αρχή, αλλά θεωρώ ότι μπορούμε να φτάσουμε σε μια συμφωνία. Δεν επιτύχαμε λοιπόν τον φιλόδοξο στόχο που είχαμε θέσει, αλλά τουλάχιστον επιτύχαμε μια συμφωνία σε ό,τι αφορά την αμοιβόμενη γονική άδεια. Η Επιτροπή αρχικά είχε προτείνει τέσσερις μήνες για τους, ε, για τους πατέρες και τις ε, μητέρες και μάλιστα πλήρη αμοιβή χωρί να υπάρχει δυνατότητα να αποζημιώνονται με άλλο τρόπο. Και τώρα έχουμε πλέον τέσσερι μήνε εκ των οποίων οι δύο όμω ε, μπορούν να εξαγοραστούν εντό εισαγωγικών, δηλαδή μπορούν να αποζημιωθούν, ενώ οι υπόλοιποι δύο είναι ε, υποχρεωτικά. Πρέπει να παραχωρηθούν από τον εργοδότη. Εμείς βέβαια είχαμε επιμείνει στο να είναι και οι τέσσερις ε, μήνες υποχρεωτικοί για τον εργοδότη. Με αυτόν τον τρόπο θέλαμε να διασφαλίσουμε τα δικαιώματα των ανδρών και των γυναικών σε ό,τι αφορά την γονική τους άδεια. Και μάλιστα να διασφαλίσουμε την ίδια άδεια για άντρες και γυναίκες. Και αυτό σε ρεαλιστική βάση, δηλαδή πραγματικά να υπάρχει ισότητα σε ό,τι αφορά αυτέ τι άδειε. Γιατί στα περισσότερα κράτη-μέλη σήμερα ε, η γονική άδεια χορηγείται στι γυναίκε κυρίω. Ε, πράγμα το οποίο βέβαια του δημιουργεί και λιγότερε δυνατότητε δραστηριοποίηση του στην αγορά εργασία. Το δικαίωμα λοιπόν γονική άδεια θα πρέπει να είναι εγγυημένο και για του άντρε και δεν θα πρέπει να είναι δυνατόν να εκχωρείται το εν λόγω δικαίωμα. Καταφέραν λοιπόν να διασφαλίσουν αυτό το δικαίωμα των ανδρών ε, παρά την ε, αντίσταση ε, που έδειξε το Συμβούλιο. Άρα λοιπόν έχουμε δύο μήνες εγγυημένης γονικής άδειας και για άνδρες και για γυναίκες. Έτσι λοιπόν διασφαλίζουμε και άδεια πατρότητας δύο μηνών πλήρως αμοιβόμενη, όπως ε, πρότεινε και η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και από εκεί και μετά έχουμε δύο συμπληρωματικούς ε, μήνες, σε ό,τι αφορά δηλαδή την ε, φροντίδα ε, του παιδιού. Όμως σε αυτή την περίπτωση τα κράτη-μέλη αποφασίζουν κατά πόσο θα είναι δυνατόν να χορηγηθεί ή όχι υποχρεωτικά από τον οικοδότη. Βέβαια το Συμβούλιο δεν ήθελε καν να υπάρξει αυτή η οδηγία και να περάσει. Οπότε το γεγονό ότι καταφέραμε έστω και έτσι να φτάσουμε σε έναν συμβιβασμό θα πρέπει να το θεωρήσουμε ω μεγάλο επίτευγμα. επιχαίρουμε το γεγονός ότι αυτή η οδηγία όχι μόνο αποτελεί εδώ ουσιαστικά την απηχή, αν θέλετε, μια κοινωνική συμφωνία στην οποία φτάσουμε, φτάνουμε, αλλά καταδεικνύει και τη μεγαλύτερη ευελιξία την οποία μπορούσαμε να δείξουμε σε θεσμικά όργανα. Ο φόβο μας ήταν ότι θα μπορούσαμε να παραβιάσουμε σε τελική ανάλυση την αρχή της επικουρικότητα. Αλλά σε τελική ανάλυση η εν λόγω οδηγία επιβεβαιώνει ότι πράγματι η κατάλληλη μορφή της ε, νομικής πράξης είναι η οδηγία. Γιατί ε, με αυτόν τον τρόπο καταφέρουμε να σεβαστούμε και τις ισχύουσε διατάξεις που ισχύουν στις ε, αγορές εργασίας των κρατών μελών. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν σε αυτές τις διαπραγματεύσεις, οι οποίες ήταν πολύ δύσκολες. Πραγματικά όλοι κατέδειξαν εδώ μια ανοιχτή και διαλλακτική στάση και έτσι καταφέραμε όλοι να εστιάσουμε στον βασικό στόχο που είχαμε θέσει εδώ. αποτελεί λοιπόν ένα μεγάλο βήμα και μια μεγάλη ε, μεταβολή και πρόοδο σε ό,τι αφορά ε, το νομικό μας ε, πλαίσιο, αυτή η νέα οδηγία. Υπάρχουν έξι κράτη-μέλη, για παράδειγμα, για τα οποία δεν προβλεπόταν καμία αποζημίωση για τη γονική άδεια. Και το ότι καταφέρνουμε εδώ να έχουμε δηλαδή τέσσερι μήνες γονική άδεια και για άνδρες και για γυναίκε είναι ένα μεγάλο επίτευγμα και επίση άδεια πατρότητα, δηλαδή γονιά, διαγιά ε, ε, δεν προβλεπόταν σε πολλές νομοθεσίες, σε πολλά κράτη-μέλη και σίγουρα δεν προβλεπόταν να είναι και αμοιβόμενο. Άρα λοιπόν, ε, είναι μια μεγάλη πρόοδος αυτή. Με αυτόν τον τρόπο περιλαμβάνουμε, αν θέλετε, και τους ε, άνδρες στην φροντίδα του παιδιού τους. Και ο η εν λόγω γονική άδεια θα πρέπει να χορηγείται ισορροπημένα και δίκαια ανάμεσα στου δύο γονεί. Η εν λόγω δηλαδή ισορροπία μεταξύ επαγγελματική και ιδιωτική ζωή αφορά και άνδρε και γυναίκε. Δεν θα πρέπει δηλαδή να είναι υποχρεωμένε οι γυναίκε να επιλέξουν ανάμεσα στο να παραμείνουν στο σπίτι ή να ε, συνεχίσουν να εργάζονται. Δεν θα πρέπει δηλαδή να είναι υποχρεωμένε να κάνουν μια τέτοια επιλογή. Θα πρέπει να συνεχίσουν να έχουν τη δυνατότητα να είναι καλέ μητέρες και τα ε, παιδιά να λαμβάνουν την φροντίδα που τους αναλογεί από τους γονείς τους και όχι από οποιονδήποτε άλλον. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο αποβαίνει προς όφελος τόσο και των δύο γονέων όσο και των παιδιών. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Αγνιέσκα, νομίζω πως ε, πραγματικά ήταν πολύ καλή δουλειά αυτή που έκανες. Ε, Μαρία Ρένα έχει τώρα το λόγο και συνέχεια ο κύριος Αγγέλκη. Μην ξεχνάτε όμω ότι έχουμε μόνο 15 λεπτά ακόμα στη διαθέση μα. Ευχαριστώ, δεν θα μακρηγορήσω. Να ευχαριστήσω την κυρία Ράγεβιτ. Ε, το θέμα είναι να βλέπουμε το ποτήρι μισοάδια μισογεμάτο. Γιατί είναι σίγουρο ότι σε σχέση με την πρόταση που είχε διατυπώσει το Ευρωκοινοβούλιο, δεν τα καταφέραμε και όλα, αλλά αυτό είναι και θέμα της έκφρασης των διαπραγματεύσεων. Νομίζω ότι αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι παρόλα αυτά πήραμε μια ρήτρα αναθεώρηση. Έτσι θα μπορέσουμε να το ξαναδούμε κάποια στιγμή με ένα νέο γύρο διαπραγματεύσεων και να ξαναδούμε όσα συμφωνήθηκαν. Είναι κάτι που μπορούμε να το επιχειρήσουμε. Όπως είπατε, είναι μια πρόοδο για την ε, άδεια πατρότητας. Εδώ όμω είμαστε στην Επιτροπή Γυναικών. Το να προβλέψουμε άδεια πατρότητας βελτιώνει την εξισορρόπηση επαγγελματικού και οικογενειακού βίου των οικογενειών. Και οι οικογένειε για μα αποτελούνται από γονεί. Ήταν σημαντικό λοιπόν να δώσουμε ένα δικαίωμα στους γονεί από την σκοπιά της άδεια πατρότητας. Όταν μιλάμε για γονεί, εννοούμε πολλέ φορές γονεί και του ιδίου φίλου. Όταν το κράτος μέλος έχει αναγνωρίσει την ομόφιλη γονεϊκότητα. Έτσι λοιπόν είναι σημαντικό να υπάρχει το δικαίωμα αυτό για τους γονείς του ίδιου φίλου και ε, μιλάμε για μέρες που αμείβονται στην περίπτωση της ε, νερωτικής άδειας. Υπάρχει μια διακριτική μεταχείριση για τις γονικές άδειες που καλύπτεται. Είναι σημαντικό λοιπόν να μην υπάρχει διάκριση ως προς την γονική άδεια θέλαμε να, να υπάρχει καλύτερη καταγραφή των δικαιωμάτων για τους γονείς και να υπάρχει δυνατότητα μη μεταφοράς για τέσσερις μήνες. Περιορίστηκε στους δύο τώρα και όχι τέσσερις. Αλλά και πάλι έχουμε τη να αναθεώρηση που θα επιτρέψει τη στιγμή που θα χρειαστεί να το ξαναδούμε και να αυξήσουμε τη διάρκεια της μη δυνατότητας μεταφοράς. Και για την άδεια, τη γονική άδεια, καταφέραμε να ξαναδούμε το επίπεδο αμοιβή, κάλυψης. Ήταν αδύνατο να έχουμε ένα σταθερό επίπεδο. Μπορέσαμε όμως να, να πετύχουμε μια μνήα μία στο επίπεδο τη ε, αμοιβή, ώστε να μπορούν τα κρατη μέλη να το επεξεργαστούν. Ένα επίπεδο που να είναι εξωπρεπέ. Κατάλληλο. ώστε οι γονεί να μην γίνουν φτωχοί, άμα γεννήσουν. Υπάρχει και μια άλλη διάσταση που προβλέφθηκε, η ρήτρα Πασαρέλα, όπως λέγεται, για κράτη-μέλη που είναι πιο γενναιόδωρα σε θέματα γονικής άδειας. όταν ξεπερνάτε ο ευρωπαϊκός μέσος Και μετά υπάρχει και μια πρόοδος για τις υπηρεσίες των φροντιστών. ένα αίτημα που είχε διατυπωθεί εδώ, στο επίπεδο της Επιτροπής μας. Πέντε μέρες το χρόνο. Είναι σημαντικό να το λέμε. Δεν καταφέραμε και εδώ να πετύχουμε το να βετε αυτό με σταθερό ποσό, όμω θα είναι το επόμενο στάδιο που θα επιτρέψει ίσω να πάμε μακρύτερα για τα θέματα αυτά τη αμοιβή. Συμφωνώ λοιπόν απολύτως ότι είναι ένα βήμα πρόοδου και ότι μπορούμε να εκφράσουμε την ικανοποίησή μας, αλλά ότι ο αγώνας δεν τελείωσε. Εάν θέλουμε πράγματι να υπάρξει ισορρόπηση επαγγελματικού και γυναικού βιού. Οι γυναίκες ακόμη ε, πληρώνουν τις συνέπειες αυτής της έλλειψης ισορροπίας. Ελπίζουμε λοιπόν το πράγμα να αλλάξει τα επόμενα χρόνια. Εκτός μικροφώνου η Πρόεδρος. Σας ευχαριστώ. Πραγματικά είναι σημαντικό το ότι αυτό το επίδομα το αναφέρουμε και ως τέτοιο. Ε, ε, και, είναι σημαντικό το ότι και η συνάδελφος ε, Μαρία Αρένα ε, ότι δηλαδή έχουμε να κάνουμε γονική άδεια. Δεν έχουμε να κάνουμε ούτε με άδεια πατρότητας ούτε με άδεια μητρότητας. Έχουμε να κάνουμε με γονική άδεια. Αν δεν το καταφέρουμε αυτό δεν θα δεν θα μπορέσουμε να αλλάξουμε την νοοτροπία. Γιατί εδώ το ζητούμενο δεν είναι απλώς και μόνο η ισότητα ε, μεταξύ ανδρών και γυναικών και πατέρων και μητερών, αλλά και μεταξύ εκείνων οι οποίοι έχουν παιδιά και εκείνων των ατέκνων. Ε, και Ακριβώ επειδή και το να έχει κανείς ε, παιδιά συνδέεται και με ένα υψηλότερο κίνδυνο ε, ένταση, ε, ήταν απαραίτητο αυτό να καταστεί σαφές και σε όλα τα κράτη-μέλη. Και σίγουρα είναι σημαντικό λοιπόν το ότι υπάρχει πλέον μια οδηγία η οποία θα ισχύει στα κράτη-μέλη και επί τη οποία βέβαια μπορεί να βασιστεί ένα κράτο μέλο για να νομοθετήσει υπεραιτέρω. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνουμε την ισότιμη μεταχείριση μεταξύ των ανδρών και γυναικών και των μητερών και των γυναικών γενικότερα. Γιατί όπω είπαμε το να είναι ε, μια γυναίκα μητέρα αποτελεί ένα παράγοντα ακριβώς για ε, ανισότητα μεταξύ μητερών και γυναικών αφενός, αλλά και μεταξύ γυναικών και άντρων αφετέρου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Γερκέ. Δεν ξέρω αν θέλεις να προσθέσεις κάτι, Αγνιέσκα. Ευχαριστώ. Θα ήθελα απλώς και μόνο να ευχαριστήσω για μία ακόμα φορά όλους τους ε, συναδέλφους, όχι μόνο τους και όδης αλλά και όσους ε, υπέβαλαν τις τροπολογίες τους. Ε, δηλαδή η δική μας γνωμοδότηση έλαβε πολλά επενετικά σχόλια. Ε, και θα ήθελα εδώ να ευχαριστήσω και τη δική μου εμπειρογνώμονα, γιατί χωρίς τη βοήθειά της δεν θα είχαμε καταφέρει μια τόσο καλή ποιότητα της γνωμοδότησής μας. Ευχαριστώ πολύ, λέει η Πρόεδρος. Αυτό ήταν το τελευταίο σημείο στην ημερήσια διάταξή μας για σήμερα. Μην ξεχνάτε ότι όμως Αύριο θα συνεχίσουμε τη συνεδρίασή μας στις 9 με την συνεδρίαση των συντονιστών. Και μετά στις 9.30 ε, έχουμε το δίκτυο για την ενσημάτωση της διάστασης του φύλου, ενώ στις 11 η ώρα θα έχουμε την εργασιακή και κοινωνική κατάσταση των γυναικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη σχετική ακρόαση. Σας ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ και την Γραμματεία, ευχαριστώ η Πρόεδρος και τους ε, διερμηνείς. Θα σας δω και πάλι αύριο. Καλό βράδυ σε όλους.